Okay, I will now start the meeting in Swedish. Uh, ni är hjärtligt välkomna till uh, uh, vårens sista sammanträde för... Ξεκινήσουμε στην τελευταία μας συνάντηση, στην τελευταία συνάντηση αυτής της σχολικής χρονιάς πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Όσον αφορά τα πρακτικά, δεν έχω λάβει μια παρατήρηση. Μπορώ να θεωρήσουμε λοιπόν ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη καταρχήν. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε αλλάξει λίγο τη σειρά των θεμάτων. Η βία κατά των γυναικών μετά από αίτημα της συγγήτριας της κυρίας Παράνοβα έχει μετατοπιστεί. Σημείο 3. Οι συστάσεις των συντονιστών πρέπει να έχετε πάρει ένα αντίγραφο στους φακέλους σας, δεν έλαβα κανένα σχόλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτές οι συστάσεις εγκρίνονται. Σημείο 4, πρακτικά Μαΐου 12, Νοέμβριος και Φεβρουάριος και 20 Μαΐου 2013. Πρόκειται για πρακτικά τα οποία θεωρώ εγκεκριμένα, καθότι ούτε για αυτά έλαβα καμία παρατήρηση ή σχόλιο. Και τώρα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων και την παρουσίαση της Προεδρίας της Λιθουανίας. Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι σήμερα την Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας της Λιθουανίας, η οποία θα μας μιλήσει για θέματα ισότητας Είστε αρμόδια για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εργασία και εμείς θέλουμε ιδιαίτερα να σας ακούσουμε σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Λιθουανίας για θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων και ισότητας των φύλων. όχι μόνο επειδή αναλάβαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και επειδή πραγματικά θέλουμε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο να συνεισφέρουμε στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να ε, προτείνουμε μια στρατηγική για την επίλυσή τους. Είναι η πρώτη φορά που η Λιθουανία έχει την Προεδρία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη για μας και είμαστε πολύ ευτυχείς που την αναλαμβάνουμε. Την ίδια ώρα βεβαίως είναι και μια μεγάλη πολύ σημαντική πρόκληση για τη χώρα μας. Το επόμενο εξάμεινο θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε επικοδομητικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, με σκοπό να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην Προεδρία της χώρας μας συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος πραγματικά εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται για έναν σημαντικότατο ρόλο όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όσον αφορά την Προεδρία μας, εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας και θα ήθελα ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω για τις ε, συναντήσεις που <clears throat> έχετε προγραμματίσει εδώ, καθώς και για την επίσκεψή σας στην πρωτεύουσα της χώρας μας, το Βίλνιους. Ο στόχος της Προεδρίας μας είναι να συνεχίσουμε με ομαλό τρόπο και απρόσκοπτα τις προσπάθειες των προηγούμενων Προεδριών και βεβαίως θα παίξουμε ένα ρόλο διαμεσολαβητή ελπίζουμε αποτελεσματικό. Θα προσπαθήσουμε σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουμε προτεραιότητες, όπως η συνέχιση των ε, εργασιών και των προσπαθειών για να ξεπεραστούν τα οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα. Η προτεραιότητά μας είναι πραγματικά μια ανοιχτή Ευρώπη με ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε όχι μόνο μία σοβαρή και σταθερή δημοσιονομική διαχείριση, ασφάλεια, αλλά και διαφορετικού τύπου ανάπτυξη έτσι ώστε να εμβαθυνθεί η ενιαία αγορά. Στηρίζουμε τους στόχους της στρατηγικής για το 2020 και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όλα αυτά βεβαίως συνδέονται αλληλένδετα με κοινέ και ίσες ευκαιρίες καθώς και με προστασία και κοινωνική ασφάλιση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο δικός μου τομέας αρμοδιότητας στις ευκαιρίες κοινωνική ασφάλιση και ισότητα κατά τη διάρκεια της προεδρίας της χώρας μου θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο άτομο, στο άτομο σε μία αναπτυσσόμενη Ευρώπη δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες ε, για ενσωμάτωση στην αγορά απασχόλησης για νέους, για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την πραγματική ισότητα και καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα ήθελα να μιλήσω για τις προτεραιότητες μας όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων και τις ίσες και ευκαιρίες ανδρών και γυναικών συμμετοχή ίση ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς. Κάτι που συνεισφέρει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία και ανάπτυξη ένας από τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Ιδιαίτερα σε τομείς όπως η απασχόληση και η κοινωνική ενσωμάτωση. Με την Ιρλανδία και την Ελλάδα, την προηγούμενη και την επόμενη Προεδρία, υπογράψαμε την δήλωση τη διακήρυξη μάλλον, στο Δουβλίνο για την ε, καταπολέμηση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων. Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε αποτελεσματικά στην ε, οικονομική ανάπτυξη, στην ανεξαρτησία την οικονομική των γυναικών και πραγματική ισότητα των φύλων. Είμαι πεπισμένη ότι οι μέχρι τώρα επικοδομητικές αποτελεσματικές προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών που έχουν την Προεδρία θα μας επιτρέψουν να πλησιάσουμε τους στόχους μας. Η Λιθουανική Προεδρία θα συγκεντρωθεί και θα προσπαθήσει να εστιάσει στα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στον τομέα της απασχόλησης έτσι ώστε να πετύχουμε αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση και να διασφαλίσουμε την θεσμική διακυβέρνηση αλλά και την ε, πρόσβαση των θεσμικών οργάνων και των ε, αρμόδιων υπηρεσιών και θεσμών στο ε, προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Στη Λιθουανία οι μηχανισμοί των διαφόρων θεσμικών οργάνων που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών ακολουθούν συγκεκριμένη στρατηγική και στόχους. Έχουμε μια πλατφόρμα για δράση και ένα συγκεκριμένο έγγραφο που περιέχει τους στόχους μας και τους θεσμικούς μηχανισμούς για να πετύχουμε την ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι μια προϋπόθεση έτσι ώστε να υλοποιηθεί στην πράξη, όχι μόνο στην νομοθεσία, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά στην καθημερινή ζωή αυτή η ισότητα δικαιωμάτων. Βεβαίως υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την ισότητα, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κάτι που είναι μια προϋπόθεση για την καλή διακυβέρνηση. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας, οι οποίες εμπεριέχονται, όπως σας είπα, σε αυτό το έγγραφο. Επίσης θέλουμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο που επιτυγχάνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα σύμφωνα βεβαίως με προκαθορισμένους δείκτες. Η de facto ισότητα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κάτι το οποίο πρέπει να εμπεριέχεται σε μεθόδους εργασίας πολλών διαφορετικών τομέων. Θα πρέπει να υπάρχουν στόχοι μετρήσιμοι. Συντονισμός, αξιολόγηση και τα αποτελέσματα να μπορούν να είναι εμφανή και να αξιολογηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο να προωθήσουμε την συμμετοχή του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ερευνητών ειδικών στον τομέα αυτό και βεβαίως τις ενώσεις και οργανώσεις των γυναικών. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε εργαλεία για το gender mainstreaming. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει μια αξιολόγηση της συνεισφοράς ανδρών και γυναικών στην συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένας δείκτης συστημικής ισότητας ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε τους στόχους μας, την υλοποίηση των στόχων μας και να αξιολογήσουμε τη μέθοδο που εφαρμόζεται. Είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να βασιστούμε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ισότητα των Φύλων. Αυτή η έρευνα, αυτή η μελέτη μας παρέχει δείκτες βάσει των οποίων θα είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές στα θεσμικά όργανα και στους μηχανισμούς των κρατών μελών, βασιζόμενοι πάντα στα συμπεράσματα της στρατηγικής της ε, Επιτροπής. Με σκοπό πάντα να πετύχουμε μια αποτελεσματική διαχείριση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Επίσης το Συμβούλιο προτείνει κάποιους στόχους και κάποια συμπεράσματα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα παρουσιάσουμε επίσης στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για την απασχόληση και την προστασία των καταναλωτών στις 30 Σεπτεμβρίου στο Βίλνιους. Οργανώνουμε μία συνάντηση βάση της ε, πλατφόρμας ε, για δράση για την αξιολόγηση των διάφορων μηχανισμών όπου θα γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα παρουσιάσουμε τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές, τη μέθοδο και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε με αποτελεσματικότητα σε κάποιες χώρες και βεβαίως τα μέτρα για το gender mainstreaming. Θα γίνει επίσης και η παρουσίαση μιας μελέτης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Όλα αυτά θα ενσωματωθούν βεβαίως στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος θα συμμετάσχει σε αυτήν την συνάντηση, δέχτηκε την πρόσκλησή μας το Σεπτέμβριο. Επίσης, για να υπάρξει συνεχής συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Λιθουανία, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οργανώνει και μία άλλη συνάντηση στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο Βίλνιους. Η ομάδα υψηλού επίπεδου για το gender mainstreaming θα συναντηθεί τις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η οδηγία για την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Εδώ πρόκειται πραγματικά για ένα τομέα όπου η απουσία ισότητας και ίσης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών είναι εμφανής. Δεν υπάρχει κατά μέσο όρο περισσότερο από 20% εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές είτε δεν υπάρχουν είτε είναι εξαιρετικά αργές σε αυτόν τον τομέα. Όταν κοιτάξουμε βεβαίως τις γυναίκες, τα νέα κορίτσια από πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, βλέπουμε ότι ο αριθμός τους είναι εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με την εκπροσώπησή τους στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Και αυτό λοιπόν προποθέτει σημαντικά αποτελεσματικά μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον οικονομικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε λοιπόν μία οδηγία που αφορά το θέμα αυτό, ιδιαίτερα για εταιρείε και επιχειρήσεις ψαγμένες στο χρηματιστήριο και οι συζητήσεις στο Συμβούλιο έχουν ε, δείξει ότι βεβαίως οι απόψεις διήστανται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει συμφωνία στην Ευρώπη όσον αφορά την ανάγκη να βελτιωθεί η ισότητα και η ίση εκπροσώπηση ε, στον οικονομικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο και απομονωμένο όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων στα επίπεδα λήψης αποφάσεων ε, στον τομέα των επιχειρήσεων. Είναι ένα πρώτο βήμα για να φτάσουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις. Εδώ βεβαίως υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ του δικαίου των επιχειρήσεων από τη μια χώρα στην άλλη. Θα πρέπει να δούμε τι ισχύει πολύ συγκεκριμένα και ποιοι είναι οι κανόνες στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων για να βελτιώσουμε την εκπροσώπηση των φίλων σε αυτά. Η Ιρλανδία παρουσίασε την πρόοδο που επετεύχθη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας της. Και βεβαίως στόχος της Λιθουανίας είναι να βρεθεί κοινή πρόταση στο Συμβούλιο και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Από την αρχή της Προεδρίας της Λιθουανίας θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το θέμα της νομικής αφήνειας αυτής της οδηγίας εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες των εθνικών νομικών συστημάτων, κάτι που θα πρέπει να αφήσει περιθώριο και ευελιξία στα κράτη-μέλη να επιλέξουν τις επιλογές τους. Όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη να μειωθεί η βία κατά των γυναικών. Βεβαίως έχει γίνει ήδη πολύ σημαντική προσπάθεια με το πρόγραμμα Τάφνη και τις προσπάθειες να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Η οδηγία η οποία επίσης καθορίζει την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και βίας. Τέλος, όσον αφορά την συντονισμένη δράση σε εθνικό αλλά και σε άλλα επίπεδα που βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία των γυναικών, την προσαγωγή των ε, εγκληματιών και την ίδια ώρα την συντονισμένη δράση. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, υποστηρίξει την στρατηγική για την καταπολέμηση κάθε είδους βίας κατά των γυναικών, την πρόληψη της βίας αυτής και το 2015 έχει οριστεί έτος για την μηδενική ανοχή στη βία κατά των γυναικών. Τα κράτη-μέλη σαφώς και θεωρούν ότι σε πολλούς τομείς υπάρχει ανάγκη για περισσότερη δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει σε πολλές μορφές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι βεβαίως γνωστό. Η συγκεκριμένη αυτή βία κατά των γυναικών, η ενδοοικογενειακή βία, είναι κάτι που πρόσφατα παρουσιάστηκε στους δείκτες για την ισότητα μεταξύ των, ε, των φύλων και παρουσιάζεται σαν μία από τις προτεραιότητες. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να επιτευχθεί πρόεδρος. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία για τις προσπάθειές της όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας τους και στην τη 27η στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, η Κάθλιν Λίντς αναφέρθηκε στις βασικές προκλήσεις στον τομέα αυτό και στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση και την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών χρειαζόμαστε μια συντονισμένη δράση που θα καλύψει πολλούς διαφορετικούς τομείς. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική δράση, ολοκληρωμένα μέτρα για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις. Θα πρέπει επίσης να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην πρόληψη και στον ε, περιορισμό και την αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε αυτή τη βία. Στη Λιθουανία έχουμε συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχία της ε, συνάντησης ε, των Ηνωμένων Εθνών που προανέφερα. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες για να επιτευχθεί περισσότερη πρόοδος στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Την ίδια ώρα θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε άλλες προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και τον καθορισμό άλλων μορφών βίας κατά των γυναικών. Μια άλλη πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι αυτή που βασίζεται στην ίση μεταχείριση όλων των ατόμων άσχετα με τις ε, θρησκευτικές, σεξουαλικές προτιμήσεις τους. Είναι κάτι το οποίο συζητείται στο Συμβούλιο βεβαίως από το 2008, δεν είναι καινούριο θέμα. Και αυτή η οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί τμήμα της ε, δικής μας σειράς προτεραιοτήτων. Όσον αφορά τα στοιχεία που περιέχει αυτή η οδηγία, οι συζητήσεις στο Συμβούλιο είναι δύσκολες. Όχι μόνο γιατί το θέμα είναι περίπλοκο, γιατί καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, αλλά και γιατί το άρθρο 19 της συνθήκης, το οποίο είναι η νομική βάση για την πρόταση αυτή, προϋποθέτει ομοφωνία απόφασης στο Συμβούλιο. Και αυτό βεβαίως οδηγεί σε μία δυσκολία όσον αφορά την ε, εξέβρεση συμβιβασμού. Όπως ξέρετε το πρόγραμμα αυτό έχει σταματήσει, έχει εμποδιστεί, θα προσπαθήσουμε όμως να επιτύχουμε περισσότερη πρόοδο. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται στους στόχους μας. Η Ιρλανδία έκανε επίσης σημαντική πρόοδο στην ομάδα εργασίας για σημαντικές πτυχές αυτής της οδηγίας. Εμείς θα συνεχίσουμε την εργασία της Ιρλανδίας και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε καταρχήν στήριξη όσον αφορά το φάσμα της οδηγίας αλλά και τον ορισμό των διακρίσεων. Έχουμε στείλει ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο θα είναι απαραίτητο για την προετοιμασία των συζητήσεων στην ομάδα εργασίας που επεξεργάζεται την οδηγία αυτή. Προσπαθούμε επίσης να κατανοήσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίζω την σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρίες. Πρόκειται για θύματα πολλαπλών διακρίσεων, αποκλεισμός, φτώχεια και θα πρέπει να στηρίξουμε τις γυναίκες αυτές με αναπηρία έτσι ώστε να προωθήσουμε την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ιδιαίτερα σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Είναι σημαντικό για να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των ε, μητέρων με αναπηρία ή των γυναικών που έχουν ανάπηρα παιδιά και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνική ζωή. Θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία με αποτελεσματικό τρόπο για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρίες και να εγγυηθούν και να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει καταρχήν να διασφαλίσουμε ότι η προστασία των ανάπηρων γυναικών είναι εγγυημένη κατά της βίας, αλλά και να προστατεύσουμε το δικαίωμά τους ε, για μία αξιοπρεπή ε, ενσωμάτωση στην κοινωνία. Τα δικαιώματα των Ρωμά. Η Ρωμά είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό παρουσίας των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι η ένταξη των Ρωμά είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ. Λίγο πριν την έναρξη της Λιθουανικής Προεδρίας, μαζί με την έκθεση για την αξιολόγηση για την ε, στρατηγική ένταξη στον Ρωμά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε και μία πρόταση ε, για τη σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη των Ρωμά. Περιέχονται λοιπόν εκεί γενικές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για μέτρα ένταξης στον τομέα της παιδείας, ε, της υγείας, της στέγασης και της κοινωνικής ασφάλισης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική για τη βελτίωση των εθνικών στρατηγικών ένταξης για τους Ρωμά. Και είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι το έγγραφο τονίζει τα θέματα των δικαιωμάτων των γυναικών και παιδιών Ρωμά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα πιο σημαντικό ε, ε, όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης των Ρωμά στην Ευρώπη. Αναμένουμε ιδιαίτερη υποστήριξη για το θέμα αυτό ε, από πλευράς Λιθουανικής Προεδρίας και θα παρακολουθούμε αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θεματολογιό μας. Στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Δεκεμβρίου ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί και η σχετική πρόταση και ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συνεισφέρει στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ένταξης των Ρωμά στα κράτη-μέλη. Και τώρα θα ήθελα εν συντομία να περάσω σε ένα ακόμα σημαντικό θέμα, την οδηγία για την ασφάλεια και την υγεία των εγγύων γυναικών ή των γυναικών που έχουν μόλις γεννήσει ε, σε κατάσταση λοχίας ή ε, θυλασμού. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες που γίνονται προκειμένου να προωθηθεί αυτό το θέμα. Δεν αποτελεί μυστικό ότι είναι περίπλοκο το συγκεκριμένο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να κάνω έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ευελιξίας για το θέμα αυτό. Βεβαίως, αναζητούμε συνένεση βάσει της πρωτοβουλίας ε, αυτής, αλλά προς το παρόν θεωρούμε ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση από πλευρά Κοινοβουλίου ή από πλευρά Συμβουλίου, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε το θέμα πιο διεξοδικά. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να με υποστηρίξετε στο επόμενο εξάμεινο, το οποίο θα είναι γεμάτο προκλήσεις η συγκεκριμένη περίοδος θα είναι πολύ σημαντική για τη Λιθουανία, θα είναι και δύσκολη φυσικά για τη Λιθουανία και κύριε Πρόεδρε τώρα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις από τις ε, Επιτροπή Γυναικών. Να δώσω καταρχάς το λόγο στους συντονιστές. Η κυρία Γκαμπριέλ καταρχάς, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη διάρκεια της Λεθουανικής Προεδρίας και να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσίαση που πρέπει να πω ότι άπτεται πολλών από τις πτυχές που συζητάμε εμείς εδώ σήμερα και ε, παραδόξως δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτηματικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συνοψίσω τα μεγάλα ερωτηματικά τα οποία μου ήρθαν ακούγοντας την παρουσίασή σας. Καταρχάς, ε, γενικά ζητήματα. Το πρώτο θέμα το οποίο πρόσεξα είναι ότι επιμείνεται ε, πάρα πολύ σε έναν ε, αποτελεσματικό διοργανικό μηχανισμό. Ποιοι είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί και πρωτίστως πώς θα καταφέρουμε να έχουμε κατάλληλες ε, επιπτώσεις ε, μέσω αυτών των μηχανισμών ε, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, διότι αυτό αναμένουν οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιους τομείς λοιπόν κατά προτεραιότητα θα ετοιμάσετε αυτούς τους μηχανισμούς και θα τους εφαρμόσετε. Δεύτερον, είπατε ότι θα συνεχίσετε τις εργασίες για την οδηγία, για την καλύτερη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών ε, στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Αναφερθήκατε σε συνένεση εντός του Συμβουλίου, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η θέση της Λιθουανικής Προεδρίας ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξει υποχρεωτική εφαρμογή ή όχι αυτής της οδηγίας και υπό αυτή την έννοια τι θα μπορούσε να κάνει η Λιθουανική Προεδρία για να διασφαλίσει την εγκυρότητα αυτού του κειμένου. Και επίσης θα να πιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα το οποίο δεν θίξατε στην παρουσίασή σας, ε, που αφορά το gender pay gap, τη διαφορά στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, έχουμε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το φαινόμενο αυτό και αυτό που απομένει είναι να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα ώστε να πάψει να υπάρχει αυτή η διαφορά η μισθολογική. Υπάρχουν εδώ και 50 χρόνια στοιχεία. Προφανώς ε, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά τα μέτρα τα οποία έχουμε εφαρμόσει και η έκθεση ε, της συναδέλφου Edith Bauer έδωσε κάποιες συστάσεις. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η έκθεση και θεωρώ ότι η Λιθουανική Προεδρία θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο θέμα αυτό και να αποτελέσει το θέμα αυτό προτεραιότητα. Διότι αναφερθήκατε στο ρόλο των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούμε να προωθήσουμε την οικονομική συμμετοχή των γυναικών και να τους δίνουμε κίνητρα για να εργαστούν όταν γνωρίζουν ότι θα ε, εξοικονομούν λιγότερα από έναν άνδρα για την ίδια θέση εργασίας και τα ίδια προσόντα. Και ένα τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να θέσω. Ε, υπάρχει κάποιο πιο συγκεκριμένο μέτρο για την υπογραφή και την κύρωση από πλευρά κρατών μελών ε, τη σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Τι θα κάνει η Λιθουανική Προεδρία για να προωθήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και πώς θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τις εθνικές πολιτικές μέσω ευρωπαϊκών μέτρων. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία πτυχή που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τον υπόλοιπο κόσμο στην εξωτερική μας δράση και στην πολιτική ανάπτυξη, αλλά και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, θα πρέπει να είναι αδιάλακτη στο θέμα της κακομεταχείρισης των γυναικών και να μην δέχεται να υπογράφει ε, συμφωνίες με χώρες εταίρους, αν δεν υπάρχει σεβασμός μεταξύ ανδρών και γυναικών και κυρίως τη βία κατά των γυναικών στις ενόπλες σειράξεις. Ε, είχα επιμείνει με την Ιρλανδική Προεδρία και ελπίζω και εσείς να κάνετε το ίδιο, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι απτά παραδείγματα στην πραγματικότητα, τα βλέπουμε καθημερινά και δεν αναφέρομαι μόνο στην περιοχή του Σαχέλ και αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Μαλί. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμψεν τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Είχα τη χαρά να σας συναντήσω στο Βίλνιους, όπου είχαμε πάει με την αντιπροσωπεία μας και ήδη από τότε ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ για την ε, Λιθουανική Προεδρία και να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει το εύρος των δραστηριοτήτων που θα αναλάβετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα που αφορούν τις γυναίκες. Αναφέρατε τη βία, αναφέρατε το mainstreaming και την ένταξη των Ρωμά. Εδώ σε αυτή την Επιτροπή έχουμε μία έκθεση για τις γυναίκες Ρωμά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και χρειαζόμαστε πραγματικά μία στρατηγική για τους Ρωμά. Γιατί παράδειγμα, για παράδειγμα στη χώρα μου οι πολιτικοί και οι πολίτες αισθάνονται πραγματικά χαμένοι όσον αφορά το πρόβλημα με τους Ρωμά. Δεν έχουν καθόλου εμπειρία, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια στρατηγική στην Ευρώπη για το πώς να χειριστούμε το πρόβλημα αυτό. Επίσης αναφερθήκατε στην οδηγία την οποία επεξεργαζόμαστε τώρα για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Θα ήθελα να μάθω πώς, ε, τι γνώμη έχετε για την ολοκλήρωση της οδηγίας κατά τη διάρκεια της Ελιθουανικής Προεδρίας. Και επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε για την οδηγία κατά των διακρίσεων. Αυτή η οδηγία έχει, περνάει από τη μία προεδρία στην άλλη. και για αυτές ε, τις ομάδες που ε, υφίστανται διακρίσεις έξω από την αγορά εργασίας. Και εδώ σε αυτή την Επιτροπή δεν ασχολούμαστε μόνο με τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και με θέματα ισότητας. Και Ορισμένες χώρες έχουν προβλήματα, για παράδειγμα με, με τους ε, ΛΟΑΔ. Πριν από λίγες εβδομάδες το Δημαρχείο του ε, Βίλνιους ε, απέριψε, αρνήθηκε να δώσει άδεια για μια διαδήλωση των ΛΟΑΔ. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η άποψή σας μάλιστα στα πλαίσια αυτής της οδηγίας κατά των διακρίσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα τα υπόλοιπα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν. Η κυρία Λινκεβίσιου τα έχει το λόγο πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Υπουργό που ήρθε στην Επιτροπή μας. Ξέρω πως αυτό δεν είναι εύκολο διότι πρέπει να συμμετέχετε σε συνεδριάσεις τριών επιτροπών και παρουσιάσατε με επιτυχία τις προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας σε άλλες δύο επιτροπές απασχόλησης κοινωνικών υποθέσεων. Η συνάδελφός μου, κυρία Τόμσον, ανέφερε πολύ σωστά ότι το πεδίο, το εύρος της Λιθουανικής ε, σειράς προτεραιοτήτων είναι μεγάλο. Αυτό που εγώ θα επιθυμούσα είναι εσείς να έχετε πραγματικά απτά αποτελέσματα τους επόμενους έξι μήνες. Θα ήθελα επίσης να πω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι η λιθουανική κυβέρνηση στηρίζει δύο πολύ σημαντικές οδηγίες. Η οδηγία κατά των διακρίσεων και εκείνη για την ε, ίση εκπροσώπηση των φέλιων στα διοικητικά συμβούλια είναι πολύ σημαντικό για την ε, Προεδρία να στηρίξει αυτές τις οδηγίες και να βρει πώς θα προχωρήσουν έτσι ώστε να ηγηθεί ενεργών διαπραγματεύσεων με τις άλλες αντιπροσωπείες. Αυτές οι δύο οδηγίες είναι αρκετά δύσκολες ως προς την επίτευξη σωστών αποτελεσμάτων και ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένοι που δεν στηρίζουν αυτές τις οδηγίες. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν εσείς αναμένετε να υπάρξει πρόοδος ε, σε αυτές τις δύο οδηγίες κατά των διακρίσεων και των, ε, της ίσης εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια. Η τελευταία οδηγία επίσης ε, εξαρτάται από το εάν εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα καταφέρουμε να βρούμε μια γρήγορη λύση. Και κάτι άλλο. Πώς είναι η συνεργασία σας με το Ινστιτούτο των δύο που εδρεύει στο Βίλνιους και τα άλλα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τις μελέτες που εκπονούνται από το Ινστιτούτο αυτό. Θεωρείτε πως η συνεργασία είναι αποτελεσματική ή μπορεί επίσης να ενισχυθεί ενδεχομένως, έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία κρατών μελών και Ινστιτούτου. Και κάτι άλλο ακόμα αναφέρατε ότι ένας από τους στόχους σας είναι η βελτίωση των ε, θεσμικών μηχανισμών. Να επαναλάβω την ερώτηση της συναδέλφου μου και εγώ. Ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα προτείνετε στο Συμβούλιο των Υπουργών έτσι ώστε αυτοί οι μηχανισμοί να έχουν αποτελέσματα, διότι υπάρχει μια αποδυνάμωση σε ορισμένα κράτη-μέλη λόγω της οικονομικής κρίσης. Σας εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ για τους ε, συντηρητικούς, ε, κύριε Γιακαντάκης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω πως με ξεχάσατε. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Υπουργό για την εξαιρετική της παρουσίαση. Είναι πάντα πολύ ευχάριστο όταν κάποιο μικρό κρατομέλος ε, αναλαμβάνει την Προεδρία, διότι είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται πόσο δημοκρατική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο ίσοι είμαστε όλοι. Η ομιλία σας ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαι σίγουρη ότι θα ηγηθείτε της Προεδρίας με δύναμη. Έχετε μεγάλες προκλήσεις. Μία από αυτές είναι και οι ποσοστώσεις και εγώ προσωπικά το ξέρετε όλοι είμαι κατά των ποσοστώσεων για πολλούς λόγους η συζήτηση θα περιστραφεί γύρω από το αν οι ποσοστώσεις θα είναι υποχρεωτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, στις 18 Σεπτεμβρίου υπάρχει μια εναλλακτική συζήτηση με τίτλο «Golden Skirts, χρυσές φούστες». Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω εκεί. Εκεί θα συζητηθεί για το αν θα μπορούν να εφαρμοστούν προαιρετικά μέτρα. Επίσης, μιλήσατε για τη βία κατά των γυναικών, το οποίο είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Η καλύτερη προσέγγιση είναι η μηδενική ανοχή. Δεν νομίζω όμως ότι αναφέρατε μία ιδιαίτερη μορφή βίας που είναι πάρα πολύ σημαντική σε πολλά κράτη-μέλη είναι ο ακροτηριασμός των ε, γεννητικών οργάνων, των εξωτερικών γεννητικών οργάνων. Εκτιμάται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 64.000 κορίτσια υφίστανται σε αυτό το μαρτύριο και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι πολλά, έχουμε πολλά να μάθουμε από τα κράτη-μέλη και να ανταλλάξουμε ε, πρακτικές με, το, με, το, με τη Γαλλία, με τις χώρες για παράδειγμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πού βρίσκεστε σχετικά με αυτό. Επίσης, αναφερθήκατε στην διακίνηση ανθρώπων. Ε, πιστεύω πως είναι ένα σημαντικό θέμα θα επιδεινωθεί η κατάσταση καθώς επιδεινώνεται και η κρίση και πιστεύω πως εμείς πρέπει να είμαστε ε, προορατικοί και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις πριν αυτές έρθουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μόρεν Σαρτιέ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω τρεις ερωτήσεις προς την Υπουργό. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την παρέμβασή σας πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτη ερώτηση όσον αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών. Μιλήσατε για τη δέσμευσή σας όσον αφορά την επίτευξη ίσων αμοιβών για τους άνδρες και τις γυναίκες. Και ακούσαμε επίσης ότι σύμφωνα με την έκθεση της Edith Bauer το θέμα αυτό μας κινητοποιεί επίσης. Πιστεύω ότι για να φτάσουμε στην ισότητα αποδοχών είναι να περάσουμε από ίσες σταδιοδρομίες. Υπάρχει μεγάλη ανισότητα στις σταδιοδρομίες ανδρών και γυναικών. Αυτή η ανισότητα στις σταδιοδρομίες ουσιαστικά οδηγεί στην ανισότητα των αμοιβών. Και την ίδια ώρα οδηγεί σε μια πολύ δυσχερή κατάσταση όταν οι γυναίκες φτάσουν στο όριο της, στην ηλικία της συνταξιοδότησης. Εκεί λοιπόν πρέπει να κινητοποιηθούμε πολιτικά για να βρούμε τρόπους να ξεπεραστεί αυτή η ανισορροπία και ανισότητα στη σταδιοδρομία ανδρών και γυναικών. Δεύτερον, σε περίοδο οικονομικής κρίσης οι μελέτες δείχνουν ότι η κρίση πλήττει πιο βία τις γυναίκες από τους άντρες. Την απασχόληση των γυναικών πλήττεται περισσότερο από αυτή των ανδρών. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να κινητοποιηθούμε και σε αυτό το σημείο. Η οικονομική κρίση ουσιαστικά είχε σαν αποτέλεσμα την απόσυρση πολλών γυναικών από μόνες τους αποχώρησαν από την αγορά απασχόλησης την αμοιβόμενη απασχόληση. Εδώ λοιπόν αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Εγώ προσπάθησα να εξετάσω τον αντίκτυπο της κρίσης επί της απασχόλησης των γυναικών και θεωρώ ότι είναι τρομερή η κατάσταση και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανισορροπία στον τομέα αυτό μετά την κρίση. Το 2014 Ζητήσαμε να χαρακτηριστεί έτος της ε, λήψης υπόψη της οικογενειακής και επαγγελματική ζωής για τις γυναίκες. Να μπει αυτό στο επίκεντρο του 2014. Είμαι εισηγήτρια, αυτό είναι το τρίτο μου σημείο, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρόκειται για ένα ταμείο που προωθεί την ε, επαγγελματική ενσωμάτωση, όπως ξέρετε, και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την ισότητα ανδρών και γυναικών, ιδιαίτερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Όλες οι πολιτικές ομάδες κινητοποιούνται στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε 25% των κονδυλίων συνοχής να ενσωματωθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να στηρίξουμε τον κοινωνικό πυλώνα της ισότητας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ακόμα ομιλητέ, ε, τρία λεπτά ο καθένας, η κυρία Γκουρμάη καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήμουν η τυχερή, συνόδευσα τον πρόεδρο όταν επισκέφθηκε την Υπουργό στη Λιθουανία και ήδη μπόρεσα να εκτιμήσω εκ των προτέρων πόσο δεσμευμένοι είστε για την υπόθεση και φυσικά και την ομάδα σα, ε, διότι πάντα χρειάζεται μια καλή ομάδα για να μα προετοιμάζει. Η Λιθουανική Προεδρία θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την ισότητα των φύλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ισότητα των φύλων ε, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα εν μέσω κρίση και θα ήθελα να πω ότι η Ελιζαμπέτ έκανε μια εξαιρετική έκθεση για τις γυναίκες εν μέσω κρίσης, παρακολούθησα τα πράγματα στενά ως και και όντως αυτή είναι μια κρίση η οποία είναι ε, ε, υφέρπουσα για τις ε, γυναίκες, διότι πλέον δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σπίτι τους να λένε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Οι γυναίκες λοιπόν ξεχάστηκαν και είναι μια χαμένη ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των γυναικών. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε πριν το τέλος της θητείας. Ε, το νομοθετικό βέβαια ε, πακέτο μέτρων που ανέλαβε η γαλλική κυβέρνηση αποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια διάθεση και ε, η παρούσα κρίση σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε θέματα ισότητας των φύλων. Εάν δεν λαμβάνουμε υπόψη τα θέματα αυτά θα έχουμε περισσότερες φτωχές γυναίκες στο μέλλον. Και φυσικά η κρίση ε, ζητά περισσότερη ισότητα, όπως είπα, περισσότερο δημοκρατική ε, για κοινωνικούς λόγους ε, και οικονομικούς λόγους. Αναφερθήκατε στην Υπουργική Διάσκεψη. Θα ήθελα κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Βέβαια ξέρω ότι θα είναι εκεί και ο πρόεδρός μας, αλλά θα ήθελα να μου διευκρινίσετε κάποια πράγματα επί του ζητήματος και ποια θα είναι η προτεραιότητα. Και θεωρώ διότι αν δεν κάνω λάθος θα υπάρξει και μία διάσκεψη για τη Μεσόγειο, για την ενδυνάμωση των γυναικών στο Παρίσι. Ε, ε, είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε κάποια πράγματα και γι' αυτό. Θα παρακολουθήσουμε στενά βεβαίως τι θα κάνετε το επόμενο εξάμενο και θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία. Δύο πραγματάκια ακόμα. Αναφερθήκατε στις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Οκτώ υπουργοί δεν ήθελαν να υπογράψουν. Αυτό αποδεικνύει ότι εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίσαμε ότι είναι πάρα πολύ σαφές ότι πρέπει ε, να επενδύσουμε σε αυτό γιατί πραγματικά θα αποκομίσουμε ωφέλη και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήθελαν να υπογράψουν. Χρειάζεστε λοιπόν μια στρατηγική για να πείσετε αυτούς τους 8 άνδρες υπουργέ οι οποίοι δεν θέλησαν να υπογράψουν και να γίνουν μέλος αυτού του εκλεκτού κλαμπ. Ε, ξέρετε ότι ε, σε κάποια κράτη-μέλη σοσιαλιστές είναι αντιπολίτευση πώς μπορούμε να έχουμε την κατάλληλη ισορροπία, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την κρίση. Και θα ήθελα να επισημάνω και εγώ αυτό που είπε η Γκαπριέλα. Υπάρχει σήμερα ένα ψήφισμα για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου και είναι πολύ σημαντική η σχέση και με την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν, όπως αναφέρθηκε, είναι διπλάσιο το πρόβλημα και εξακολουθεί να στέλνει γυναίκες ε, προς τη φτώχεια. Και τέλος η οδηγία για τη μητρότητα. Είχαμε την εξαιρετική αντιπρόεδρο την κυρία Στρέλα που ασχολήθηκε με το θέμα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και είναι πονίδιστο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να προχωρήσει το θέμα προαιρετέρω. Ευχαριστώ. Η κυρία Στρέλα είναι η τελευταία στον κατάλογο των μιλητών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω την Υπουργό. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την παρουσίασή της και να της ευχηθώ καλή επιτυχία για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο μας παρουσίασε. Η ερώτησή μου αφορά την αναθεώρηση της λεγόμενης οδηγίας για την άδεια μητρότητας η οποία δυστυχώς ε, βρίσκεται σε τέλμα στο Συμβούλιο από τον Οκτώβριο του 2010. Εντός ολίγου θα έχουμε ευρωεκλογέ ε, του χρόνου το Μάιο πιο συγκεκριμένα και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να γίνει κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρούμε ότι πρέπει να δράσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Πολλό μάλλον, διότι αν δεν κάνουμε τίποτα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι για πέντε χρόνια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό για τις ευρωπαϊκές οικογένειες. σε μια χρονική συγκυρία στην οποία η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είναι σε ανησυχητικά ποσοστά, είναι τόσο χαμηλά δηλαδή τα ποσοστά, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα προκειμένου οι πολίτες να μπορέσουν να συνεχίσουν να μας εμπιστεύονται. Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον ε, υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις ε, για να εκμεταλλευτούμε τις προσπάθειες που έκανε ε, και η Ιρλανδική Προεδρία αλλά και οι προσπάθειες ε, που έκανε η αρμόδια υπουργό και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Υπουργό Κάθλιν Λίντς ε, για τη δέσμευση που επέδειξε, διότι πραγματικά έκανε μία απόπειρα να ξεμπλοκάρει αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο. Τώρα, η κρίση πολλές φορές αποτελεί άλοθη για να γίνονται λιγότερες επενδύσεις στις κοινωνικές πολιτικές. Αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό από την οικονομική ε, κρίση. Η συγκεκριμένη οδηγία εντάσσεται σε ένα σύνολο μέτρων που στόχο έχουν να αναστρέψουν αυτή τη δημοκρατική τάση η οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Υπάρχουν ε, εμπειρογνώμονες θέματα δημογραφίας ε, που επιμένουν στο γεγονός ότι αν δεν αναστραφεί αυτή η πτωτική τάση, η Ευρώπη όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς ε, σήμερα θα πάψει να εφίσταται η γυράσκουσα κοινωνία, το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων, όλα αυτά αναδιαμορφώνουν τον πληθυσμό της Ευρώπης. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτό υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι ε, αρκετές φορές ε, φάνηκε ότι υπάρχει ευελιξία από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι διατεθειμένο να συζητήσει. Ελπίζω το Συμβούλιο να κάνει και αυτό ό,τι το αναλογεί. Δηλαδή, να κάνει το αποφασιστικό βήμα, να συνεισφέρει προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μια συμφωνία η οποία θα είναι ανάλογη των, προσδιοκών και, των προσδοκιών και των ευαισθησιών των ε, οικογενειών της Ευρώπης. Εάν δεν ξεκινήσει έστω ένας υποδιπόδης διάλογος, θα είναι αδύνατον να δούμε πού υπάρχουν κοινά σημεία και πού υπάρχουν αποκλήσεις. Το πλέον σημαντικό λοιπόν είναι να ξεκινήσει τουλάχιστον ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και ε, θα δούμε τι μελιγενέστε. Από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε μεγάλη διάθεση ευελιξίας ακριβώς για να καταλήξουμε σε μια λύση. Ελπίζω το Συμβούλιο να αποστείλει το ίδιο μήνυμα ευελιξίας και διάθεσης προς συζήτηση. Ε, κυρία Υπουργέ, όχι μόνο εγώ αλλά και οι συνάδελφοι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό από τις αρχές του 2009 και ε, ασχοληθήκαμε με το θέμα με όλες τις εκπεριτροπής Προεδρίας και από πλευρά Συμβουλίου η απάντηση ήταν συνεχώς μηδέν. Το απόλυτο μηδέν, συνεχής απογοήτευση. του χρόνου θα έχουμε προεκλογική εκστρατεία και πολλές κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εξηγήσουν στις οικογένειες και στις ε, γυναίκες της Ευρώπης γιατί δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν έστω ένα διάλογο. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να εγκριθεί ε, οπωσδήποτε η πρόταση, δεν λέω ότι θα πρέπει να εγκριθούν τα μέτρα τα οποία ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν υπήρξε καν μία χειρονομία ε, ως ένδειξη σεβασμού και διάθεσης για διάλογο με τους... Ε, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο Υπουργός θα απαντήσει στα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ξέρω ότι ήταν πολλέ οι ερωτήσεις και πολλά τα σχόλια. Δυστυχώ όμω δεν έχετε πάνω από 10 λεπτά για να απαντήσετε σε όλα αυτά. Σα παρακαλώ λοιπόν, προσπαθήστε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ερωτήσεις και τις ευχές σας. Θα τα λάβουμε όλα αυτά σοβαρά υπόψη μας τους επόμενους έξι μήνες. Κύριε Πρόεδρε, σωστά είπατε ότι οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές, προσπάθησα να τις σημειώσω. Οι ερωτήσεις αυτές και τα σχόλια θα μας βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε τη δουλειά μας. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τουλάχιστον ε, μία ερώτηση κάθε μέλους. Καταρχάς, κυρία Γκάμπριελ, ε, μιλήσατε για ποσοστώσεις και για εις εκπροσώπηση και ποια είναι η θέση της ε, Λιθουανικής Προεδρίας σε αυτό. Όπως ανέφερα, Θα δώσουμε έμφαση στην πρωτοβουλία αυτή. Θα είναι μία από τις κυριότερες προτεραιότητές μας. Και στην ατζέντα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ. Ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε πρόοδο. Ξέρουμε πως είναι κάτι το δύσκολο διότι κάθε κράτος μέλος έχει την δική του αφετηρία στις διαπραγματεύσεις. Η κατάσταση είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα, οι απόψεις διαφέρουν πολύ. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε νομική σαφήνεια και αναλογικότητα στις διατάξεις του της οδηγίας. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι ο στόχος ε, της ε, οδηγίας θα είναι όσο το δυνατόν σαφέστερος, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μην έχουν ερωτήσεις όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας, ε, οι οποίες θα είναι περιττές. Αναφέρεται επίσης στην σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η Λιθουανία έχει υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Αναφέρεται επίσης το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που επιμένει, που παραμένει. Και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να εξαλειφθεί αυτό το μισθολογικό χάσμα. Υπάρχει βέβαια μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των άνθρωπων ε, από χώρα σε χώρα και αυτό το πρόβλημα πλήττει τις γυναίκες ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών. Και αυτό το ζήτημα λοιπόν χρειάζεται την άμεση προσοχή μας. Τώρα, θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Τόμσον. Ρωτήσατε για πολύ σχετικά ζητήματα με αυτά που κάνουμε. Για παράδειγμα, για την κατάσταση των Ρωμά. Αναφέρατε επίσης την ένταξη των γυναικών Ρωμά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Και τώρα όσον αφορά την ε, οδηγία για την ε, για κατά των διακρίσεων, να σας πω ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Το άρθρο 19 προϋποθέτει ομοφωνία στο Συμβούλιο και εδώ βρίσκεται και η αιτία των συγκρούσεων, εδώ βρίσκεται και η αιτία που, έχει, που έχουν μπλοκαριστεί διαπραγματεύσεις. Τώρα όσον αφορά τους ΛΟΑΔ και το συμβάν στο Βίλνιους, να σας πω ότι το φεστιβάλ υπερηφάνειας, η παρέλαση θα ε, συζητιέται πού θα λάβει χώρα, σε ποιου ε, δρόμου. Η συνάδελφος ούτε ανέφερε επίσης το Ινστιτούτο Ισότητας και μας έκανε ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Χαιρόμαστε πολύ για την συνεργασία που έχουμε με το Ινστιτούτο. Όλα τα κρατημέλη χρησιμοποιούν τις ε, μελέτες και τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου αυτού. Αυτές οι μελέτες που συντάσσει το το Ινστιτούτο αυτό μας βοηθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Ινστιτούτο αυτό λειτουργεί σαν ένα ίδρυμα που γίνονται εις βάθος αναλύσεις των προβλημάτων σχετικών με την ισότητα. Η κυρία Γκάμπριελ επίσης, καθώς και άλλες ευρωβουλευτές, ρώτησαν για τους ε, θεσμικούς μηχανισμούς. Αυτή είναι μια κύρια προτεραιότητά μας, βασισμένη στην πλατφόρμα του Πεκίνου, Υπάρχουν ακόμα διαφορές ε, όσον αφορά την θέση ανδρών και γυναικών. Η πρόοδος είναι αργή και χωρίς πραγματική ισότητα και πραγματικούς στόχους ισότητας είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε και τους στόχους της Ευρώπης 2020. Τώρα, όσον αφορά την απασχόληση. δεν έχουμε επιτύχει ακόμα ούτε σε επίπεδο κοινοτικό ούτε σε επίπεδο κρατών μέλων πραγματική ισότητα. Αλλά για να διασφαλίσουμε ότι δεν μένουμε μόνο στα λόγια και ότι θα υπάρχει ισότητα και στην πράξη, χρειαζόμαστε αποτελεσματική διαχείριση, διαχείριση προσανατολισμών προς αποτελέσματα στα θεσμικά όργανα και σωστούς μηχανισμούς για να έχουμε λοιπόν αυτά τα σωστά αποτελέσματα. Αυτό αναφέρεται στην πλατφόρμα του Πεκίνου και στο ε, Σύμφωνο Ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα. Ανέφερε επίσης ε, την ε, δήλωση για την ισότητα όπου αναφέρεται ότι το δυναμικό και ανδρών και γυναικών πρέπει να χρησιμοποιείται εξίσου και αυτό θα δώσει την προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη ώστε αυτά να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συνόλου της. Έχουν προταθεί λοιπόν συγκεκριμένες δράσεις στον ε, τομέα της ενίσχυσης των ε, ανθρώπινων δυνατοτήτων, της συλλογή στατιστικών στοιχείων, τα οποία θα, θα αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της ισότητας και κάτι άλλο σημαντικό όσον αφορά τους θεσμικούς μηχανισμούς είναι ότι υπάρχει ανάγκη ελέγχου και αναφοράς. Αυτά ως προς τους θεσμικούς μηχανισμούς. Τώρα θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Κοντακή. Αναφέρατε τις ποσοστώσεις στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Αναφέρατε την ευεία κατά των γυναικών. Η δική μου θέση είναι πως δεν πρέπει να υπάρχει ανοχή στη βία από που αυτή και αν προέρχεται. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς από το 2008 έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο και συνεχίζεται ακόμα διότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο πεδίο εφαρμογής των ποσοστώσεων και όχι μόνο. Και πάλι το άρθρο 19 εδώ είναι σημαντικό, διότι όπως είπα απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε ακόμα να επιτύχουμε κάποιον συμβιβασμό. Ωστόσο κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να εξαλείψουμε τη βία από τους ε, διάφορους ε, τομείς της κοινωνίας και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Θα ήθελα τώρα να απαντήσω στην κυρία Σαρτιέ. Μιλήσατε για ίσες ευκαιρίες ε, για άνδρες και γυναίκες. Για τις ανισότητες που παρατηρούνται να σας πω ότι η έλλειψη ισότητας μισθολογικής είναι κάτι το αρνητικό. Γνωρίζουμε ότι το μισθολογικό χάσμα έχει ένα ποσοστό 16,2%. Στη Λιθουανία η διαφορά είναι μικρότερη, είναι γύρω στο 12%. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα χρειάζεται μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, μία σφαιρική αντιμετώπιση. Επίσης, σημαντικό επίσης είναι οι πολίτες που φτάνουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Ορισμένοι από αυτούς απαιτούν πρόσθετες ε, υπηρεσίες και επιδοτήσεις επειδή δεν μπορούν να ζήσουν με τις συντάξεις που παίρνουν. Ε, να σας πω ότι πιστεύω πως η κρίση δεν πρέπει να είναι δικαιολογία, δεν είναι η αιτία για όλα τα προβλήματά μας. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα βρούμε διαφορετικές λύσεις μαζί. και να μην θεωρούμε την ε, κρίση ως το μόνο παράγοντα. Και κάτι άλλο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, είτε αυτό είναι, έχει ανδρικό φύλλο είτε γυναικείο, είναι εξίσου σημαντικές. Είναι σημαντικές και σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο και συνεισφέρουν οι επενδύσει αυτέ στην ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσει, επενδύσει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τώρα θα απαντήσω στην κυρία Γκουρμάη. Όπως ε, είπα και για το μισθολογικό χάσμα, πιστεύω πως αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε πρόοδο στο ζήτημα αυτό. Όπως σας είπα, σχεδιάζουμε μια εκδήλωση, μια εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στους θεσμικούς μηχανισμούς και χαίρομαι πολύ που το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων έχει δηλώσει πανέτοιμο να μας βοηθήσει, μας έχει δώσει μελέτες και πολύ υλικό για το συνέδριο αυτό. Εάν λοιπόν έχετε τον ε, χρόνο, θα ήθελα να σας καλέσω να συμμετάσχετε στο συνέδριο αυτό. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο στο Παρίσι, θα ε, προσπαθήσω να παρευρεθώ Ξέρω πώς τα θέματα αυτά είναι σημαντικά και για την Επιτροπή σας και για τα κρατημέλη. Αυτά, νομίζω. Τέλος, θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Εστρέλα για την ε, οδηγία μητρότητας. ως ε, υπουργό. Αρμόδια, πιστεύω πως όλες οι μητέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν καριέρα και οικογένεια και ανατροφή παιδιών. Ξέρω πως αυτή η οδηγία περιμητρότητας είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει μία διαμητρότητα 20 εβδομάδων με πλήρε απολαυέ κατά τη διάρκεια των 27 εβδομάδων. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία εδώ. Αλλά είμαι πεπισμένη πώς θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάποια λύση κατά τη διάρκεια της δικής μας προεδρίας. Στηρίζω όμως ε, οπωσδήποτε τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες σας. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι τα ποσοστά των ε, γεννήσεων μειώνονται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι η στάση των ανθρώπων προς τις γυναίκες, προς τις μητέρες στα κράτη-μέλη είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς λοιπόν θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να βρούμε κάποια σωστή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Βλέπετε ότι είμαστε δεσμευμένοι. Οι ερωτήσεις είναι πολλές και είμαστε πολύ ευτυχείς που μπορέσατε και ήρθατε στην αρχή της Προεδρίας σας. Αναφέρετε πολλά θέματα ενδιαφέροντα για μας, ουσιαστικά, που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεγάλο βαθμό. Σας ευχόμαστε επιτυχία για την εξάμεινη Προεδρία σας.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 συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Και έχω την ε, τιμή να σας παρουσιάσω την ε, νέα Ιταλίδα Υπουργό Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, την κυρία Σεσίλ Κιέγγε. Από τότε που αναλάβατε καθήκοντα, πρέπει να πω ότι τραβήξατε την προσοχή της Επιτρεπής μας, διότι είστε η πρώτη γυναίκα ε, μαύρη προερχόμενη από την Αφρική ε, σε μια ευρωπαϊκή χώρα που τέλει καθήκοντα υπουργό και υπάρχουν δύο εκθέσεις ε, τις οποίες εξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και έχουν άμεση σχέση με τα καθήκοντά σας. Το ένα είναι το θέμα της ένταξης στο Ρωμά και επίσης έχουμε και μία έκθεση η οποία αφορά τους μετανάστες ε, χωρίς ε, έγγραφα. Ο διορισμός σας λοιπόν πραγματικά μας ε, εντυπωσίασε, μας ενδιέφερε και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ. Και επειδή ακριβώς ήσασταν αντικείμενο αρκετών ρατσιστικών και φιλετικών επιθέσεων, ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να είμαστε εδώ σήμερα μαζί για να κάνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Να σας δώσω λοιπόν απευθεία το λόγο και στη συνέχεια θα υπάρξουν σίγουρα ερωτήσεις. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω. Grazie. Ε, ringrazio il Presidente della Commissione per eh, i diritti delle ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων για την ε, πρόσκληση που με και μπορώ να είμαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ και να ε, έχω την ευκαιρία να αναφερθώ σε κάποια θέματα ως Υπουργός ε, Ενσωμάτωσης. Η ισότητα των φύλων, επομένως και ίσες ευκαιρίες. Πρόκειται για αρχές οι οποίες σήμερα θεωρούνται εγκάρσιες, διότι άπτονται πολλών από των σημαντικών πτυχών της κοινωνίας μας. Όσον αφορά την Ιταλία, θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινίσω ότι από το 1996 δόθηκε από τις κυβερνήσεις ε, ε, κάθε φορά ε, αντίστοιχη αρμοδιότητα είτε σε Υπουργό είτε σε Γενικό Γραμματέα. Και στην Επιτροπή σας θα ήθελα να ε, σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την υποστήριξη μετά από τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο Σούλτς. Όσον αφορά τα αρμοδιότητές μου, θα ήθελα να σας πω λίγα πράγματα για το στόχο, την πρόταση και το συντονισμό των πρωτοβουλειών για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πολιτικών ισότητας και ίσων ευκαιριών οι παρεμβάσεις ε, για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις αρχές και στις διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έγκριση πρωτοβουλειών για την εκπροσώπηση της ελληνικής κυβέρνησης στις σχέσεις ε, με διεθνείς οργανισμούς η πρόβλεψη στην Ιταλική νομοθεσία ενό υπουργού ή ενό γενικού ε, γραμματέα, ο οποίος θα ασχολείται συγκεκριμένα με τα θέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο και τη σημερινή μα συνάντηση και ε, αυτό αποδεικνύει ότι είναι πολύ σημαντικά και πάντα επίκαιρα. Αλλά επίση, το γεγονός ότι έχω αναλάβει θέματα ένταξης για να ε, αντιμετωπίσω τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Καταρχάς ότι είναι εγκάρσιο αυτός ο χαρακτήρας και τα θέματα ισότητα και φύλων εξακολουθούν να είναι πάντα επίκαιρα. Και είναι προφανές ότι φαινόμενα ε, δεν, τέτοιου τύπου ε, δεν μπορούν να θεωρούνται ότι είναι αυτόνομα, αλλά θα πρέπει να τα εξετάζουμε στο σύνολό τους. Στην Ιταλία και στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια βιώνουμε μια ε, βαθιά μετάλλαξη η οποία προκύπτει από το φαινόμενο της μετανάστευσης και ε, οι χώρες μας και η Ήπειρός μας μετατρέπεται από χώρες ε, μετανάστευσης σε χώρες υποδοχής μεταναστών που σημαίνει ότι αλλάζει ε, το προφίλ και πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Στο νέο πλαίσιο οι μετανάστες είναι ε, πρωταγωνιστές πολύπλοκων δεδομένων που αφορούν την οικονομία, τον πολιτισμό, την κοινωνία στις χώρες υποδοχής και στις χώρες καταγωγής και από εκεί και πέρα επεκτείνονται και σε άλλες ε, επικράτειες η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο διαρθρωτικό στις κοινωνίες μας και μπορεί να δημιουργήσει πολύ σημαντικές ευαίσθητες αλλαγές στον κοινωνικό ιστό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, στην καθημερινή ζωή και να δεχτούμε το γεγονός ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει με ίσο και ε, αξιοπρεπή τρόπο. Αλλά για να μπορεί κάποιος να ζει με αξιοπρεπή και ισότιμο τρόπο ε, θα πρέπει να εξετάσουμε και τα δικαιώματα των γυναικών και κυρίως των γυναικών μεταναστών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω κάποιες από τις διατάξεις του Ιταλικού Συντάγματος. Το άρθρο 2, το οποίο αναγνωρίζει την ε, ε, εγγύηση στα παραβίαστα δικαιώματα του ανθρώπου και το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει πολιτική, οικονομική και κοινωνική αλληλεγγύη. Το άρθρο 3 το οποίο προβλέπει να απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση που βασίζεται σε φύλλο, ε, γλώσσα, θρησκεία, πολιτικές απόψεις, ε, προσωπικές και κοινωνικές ε, συνθήκες και αναθέτει στην Ιταλική Δημοκρατία το καθήκον να άρει οποιαδήποτε προσκόμματα οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα που περιορίζουν την ελευθερία και την ισότητα των πολιτών και δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπου και την ε, αποτελεσματική συμμετοχή ε, στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση της χώρας. Υπάρχει επίσης το άρθρο 37, το οποίο προβλέπει για την εργαζόμενη γυναίκα τα ίδια δικαιώματα και ισότιμες συνθήκες εργασίας και την ίδια μισθολογική κλίμακα με όλους τους εργαζομένους. Οι κανόνες θα πρέπει να προβλέπουν στις γυναίκες εργαζόμενες ε, την ε, ε, προσαρμογή με τα οικογενειακό της καθήκοντα και ταυτόχρονα να υπάρχει και συγκεκριμένη ασφάλιση για την προστασία της μητέρας και του παιδιού. Πρόκειται για θεμελιώδους κανόνες, οι οποίοι ε, δεν είναι μόνο θέμα αρχής, αλλά είναι και πολύ ισχυροί ως προς το περιεχόμενο τους και αφορούν ε, συμπεριφορές ε, τις οποίες πρέπει να υλοποιεί το κράτος. Βέβαια, χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να μεταφραστούν όλα αυτά σε συστατικά στοιχεία της ισότητας και των ίσων ευκαιριών. Δεν θεωρώ ότι εδώ είναι η στιγμή να αρχίσουμε να εξετάζουμε όλη την πορεία που ακολούθησε η Ιταλία για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι θα γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα. Δικαιώματα των γυναικών, στην ισότητα των φίλων και στις ίσες ευκαιρίες. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι πολλά σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν σε θέματα οικογενειακού δικαίου, βίας ε, κατά των γυναικών, πρόσβασης των γυναικών στα επαγγέλματα και στη δημόσια αξιώματα. Και φυσικά η πορεία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, όπως αποδεικνύουν και ε, κάποια στοιχεία, διότι κάποιες παρεμβάσεις, ακόμα και σε νομοθετικό επίπεδο, ε, δείχνουν ε, τι έγινε τους τελευταίους μήνες. Πρόσφατα, στις 19 Ιουνίου, το Ιταλικό Κοινοβούλιο ε, κύρωσε τη συνθήκη της ε, Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας. Η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει αμέσως να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα ε, περιστατικά αυτά και να προβλέψουν τη βία και να προστατέψουν τα θύματα. Το 2012 στην Ιταλία ε, καταγράφησαν 124 περιπτώσεις ε, δολοφονιών γυναικών και πέρσι ε, βλέπουμε ότι συμβαίνουν αντίστοιχα φαινόμενα με φέτος. Στις 30 ε, Νοεμβρίου του 2012 που αφορά, μια νομοθεσία που αφορά κανόνες για την πρόσβαση στην δημόσια διοίκηση ε, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον ενισχύει κανόνες για τις ποσοστώσεις σε θέματα φύλων. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι νέοι κανόνες υπάρχουν ποινές που προβλέπουν και την ε, ε, αναστολή λειτουργίας του κοινωνικού οργάνου και θα πρέπει να ανανεωθεί με άλλους τρόπους ε, σε συγκεκριμένες προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο. Υπάρχει άλλη πρόσφατη διάταξη, νόμος του 23 Νοεμβρίου του 2012, υπαριθμών 215, που αφορά τη νέα ισορροπία της εκπροσώπησης ε, γυναικών ε, και σε τοπικές και περιφερειακές ε, αυτοδιοικήσεις και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ε, προσώπηση και των δύο φύλων και τη δυνατότητα οι ψηφοφόροι σε δήμους ε, με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων να ψηφίζουν διπλά έναν υποψήφιο από κάθε φύλο. Όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε θέματα δικαιωμάτων των γυναικών και προστασίας των γυναικών από τη βία και αυτό σημαίνει ότι ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οποιαδήποτε σημαντική πορεία όπως ε, αυτή που αφορά τις ε, βασικές θεμελιώδεις αρχές της ε, κοινωνίας πρέπει πάντα να συνοδεύεται και από μία αλλαγή νοοτροπίας. Επίσης, μας ενδιαφέρει το θέμα των σχολείων. Στα σχολεία είναι ο χώρος συνάντησης και αντιπαράθεσης. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι στις χώρες υποδοχής η παρουσία κάποιων αλλοδαπών ε, μαθητών από διάφορα εθνικότητες έχει μια διπλή αξία. Καταρχάς, μέσω της εκμάθησης της ε, γλώσσας ε, της χώρας υποδοχής, είναι, έχουμε το εφαλτήριο αυτής της πορείας και είναι και μια ευκαιρία να μάθουν τα παιδιά και τις διάφορες γλώσσες των συμμαθητών τους, τις παραδόσεις τους και τον πολιτισμό τους η πορεία της ολοκλήρωσης είναι μακρά και περίπλοκη και σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει προσοχή ε, συνεχής ε, και ε, πέρα από το σχολείο πολύ σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν και οι πολιτιστικοί διαμεσολαβητές που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους μετανάστες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Ε, από την πρώτη στιγμή λοιπόν της άφηξης ε, στην χώρα προορισμού θα πρέπει να απευθυνθούμε στις γυναίκες διότι πρόκειται για γυναίκες οι οποίες πολλές φορές αποτέλεσαν αντικείμενα πολύ σοβαρών εκκλημάτων ε, παραδείγματος χάρη σεξουαλική εκμετάλλευση στο χώρο εργασίας, ε, ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων και για το ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στα πλαίσια της οικογένειας, την οποία προστατεύουν και προασπίζονται ανα πάσα στιγμή. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ στην ιδιαίτερη προσοχή που έδωσε η κυβέρνηση για το ένταλμα ευρωπαϊκής προστασίας για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και κάποιες περιπτώσεις προστασίας γυναικών στον ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον, άκουσα ότι είναι μεγάλο και το ενδιαφέρον σας ε, για το, ε, όσα προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο μου για το γύρο τραπέζης ε, για το θέμα αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολλά σε εθνικό επίπεδο και πραγματικά θα μπορέσω να ε, συζητήσω για τα θέματα αυτά και μαζί σας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η πλήρες επίτευξη των στόχων της ισότητας και των ίσων ευκαιριών αποτελεί ένα κοινό στόχο για όλους όσους πιστεύουν στις αξίες της δημοκρατίας. Αν όντω πρωταγωνιστή στη μάχη για την ισότητα των φίλων είναι οι γυναίκες, άλλο τόσο η σημαντική συνεισφορά των γυναικών είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δώσουν μαζί τη μάχη για να ε, κατακτήσουν ε, τη δικαιοσύνη. Και το να προχωρήσει κάποιος τη μάχη για να εγγυθούν ε, σε όλους μία αξιοπρεπή διαβίωση δεν είναι αρμοδιότητα μόνο όσων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από κοινωνική και οικονομική πλευράς δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τη συνεισφορά που θα μπορούσαν να δώσουν ε, οι κοινότητες και ο καθένας μεμονωμένα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήνουμε τη δυνατότητα να μπορεί ο καθένας να αναπτυχθεί, διότι αλλιώς θα έχουμε αρνητικές συνέπειες για την οικονομική και κοινωνική ευημερία μιας χώρας. Στην ε, πραγματικότητα λοιπόν έχουμε καταπασπατάληση ανθρωπίνων χώρων, δεδομένου δε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της ε, λόγω της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης ε, και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο να υποστεί τέτοια προβλήματα. Θα ήταν αδικία και ε, για τις θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες αναφέρθηκα. Ευχαριστώ. Thank you so much for Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη για ερωτήσεις ή σχόλια. Καταρχάς τους συντονιστές για το ΕΛ, κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Καταρχά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη σημερινή σα επίσκεψη στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Είναι χαρά να σα έχουμε εδώ. Καταρχά, διότι είστε ζωντανή εικόνα τη συμμετοχή των γυναικών ε, στο πολιτικό προσκήνιο και μάλιστα σε ένα Υπουργείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ιταλία αλλά για όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Επίση, γιατί έχετε ένα θετικό μήνυμα ανοχή και φυσικά αυτό το κάνετε με ευφυα. Βλέπουμε πώς αντιδράσατε στις ε, ρατσιστικές ε, επιθέσεις ε, τις οποίες δεχθήκατε από τότε που αναλάβατε καθήκοντα στην Ιταλική κυβέρνηση και αυτές φυσικά τις καταδικάζουμε. Αλλά οι επιθέσεις αυτές ορισμένες φορές αποτελούν και το έναυσμα για να ξεκινήσει η συζήτηση και να αντιληφθούμε ότι η ένταξη δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αγνοήσουμε πλέον, δεν μπορούν να το αγνοήσουν ούτε οι Ιταλοί ούτε οι Ευρωπαίοι και θα πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα καλύτερα στοιχεία της διαφορετικότητας ε, παντού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσίασή σας και αντιλαμβάνομαι ότι τα καθήκοντά σας είναι πολύ σημαντικά αλλά και σημαντικά ε, και για μας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο πτυχές. Αφενός, ε, συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι οι γυναίκες ε, μετανάστες θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής, διότι βρίσκονται ενώπιον διακρίσεων πολλαπλών και στη χώρα υποδοχής αλλά και στη χώρα καταγωγής τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίσουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να διευκολύνουμε την ένταξη να φτάσουμε μέχρι τις γυναίκες. Σε ατομικό επίπεδο και οι γυναίκες οι οποίες έχουν μία εξειδίκευση, κάποιες δεξιότητες και προσόντα να αναγνωρίζονται αυτά, αν είναι μετανάστες, να μην παραμένουν εξαρτώμενες στη χώρα υποδοχής. Θα πρέπει επίσης να δούμε και την προστασία των γυναικών που δεν έχουν ε, ειδίκευση, διότι απειλούνται και μπορούν να γίνουν θύματα λαθρεμπορίου. Βεβαίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά απασχόλησης και για τις δύο αυτές κατηγορίες γυναικών υπάρχουν ακόμα πολλές δυσκολίες και εμπόδια. Δεύτερον, αναφερθήκατε στη βία κατά των γυναικών και εμείς σας ενθαρρύνουμε, σας στηρίζουμε έτσι ώστε το κράτος από το οποίο προέρχεστε να τροποποιήσει την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε πώς με εκστρατείες ευαισθητοποίησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει σεβασμός των γυναικών και προστασία των δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά τις εκλογές στην η Δημοκρατία του Κονγκό, Κυρία Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι για όλες τις γυναίκες που ζουν σε αυτή τη χώρα, οι οποίες βεβαίως είναι δυνατές αλλά χρειάζονται την υποστήριξή μας, είστε μια σημαντική ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Στις 11 πρέπει να αρχίσει η ψηφοφορία. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν όταν παίρνετε το λόγο να είστε σύντομοι. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την Υπουργό και νομίζω ότι όχι μόνο ως Ευρωβουλευτής αλλά και ως γυναίκα εκφράζω την απόλυτη ακονοποίησή μου για αυτή την τόσο σημαντική επιλογή που έκανε ο Πρωθυπουργό Λέτα και για πρώτη φορά έδωσε υπουργικό θόκο σε μια Ιταλίδα πολίτη που γεννήθηκε στην Αφρική. Και νομίζω ότι αυτό αυτό το γνωρίζουν οι συνάδελφοι και αποτελεί συμβολικ... κίνηση συμβολικού χαρακτήρα και στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα διότι συνδυάσατε πάρα πολύ καλά τα ισότητα των γυναικών και τις ίσες ευκαιρίες με το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι ε, εγγεγραμμένα όλα αυτά σε πολιτικές μετανάστευσης και δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τις γυναίκες μετανάστρες, διότι αυτές είναι το βασικό αντικείμενο της ένταξης. Πολλές φορές οι γυναίκες, ακόμα και στη χώρα μας, είναι πολύ πιο ήρεμες και πολύ πιο αποτελεσματικές, διότι οι γυναίκες αποτελούν το ισχυρό στοιχείο της ενσωμάτωσης και νομίζω ότι και η προσωπική σας ιστορία το αποδεικνύει. Γνωρίζω επίσης ότι θέλετε να ασχοληθείτε με διάφορα μέτωπα σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία και θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθείτε και με το συμβολικό χαρακτήρα της κατάλληλης επικοινωνίας. Οι επιθέσεις ε, που υπήρξαν και εδώ στο Κοινοβούλιο και χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που ο Υπουργό είπε ότι στην βία θέλει να απαντήσει στο μέγιστο βαθμό με την αντίθετη πτυχή χωρίς καθόλου βία και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει όχι μόνο σε κάποια περιθωριοποιημένα ε, τμήματα της κοινωνίας αλλά και στα πιο ε, ανώτερα στρώματα, πιο μορφωμένα, να μην υπάρχει ξενοφοβία και να μην ε, ε, θεωρείται ότι είναι πολιτιστικό πρόβλημα το θέμα της συμβίωσης. Μου άρεσε επίσης ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπατε για τη διάθεση της Ιταλίας να εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές διατάξεις και φυσικά την παραπομπή που κάνατε στην οδηγία για την εμπορία ανθρώπων, που είναι κάτι ε, ε, για το οποίο βέβαια η Ιταλία έχει αρκετά προχωρημένη νομοθεσία. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς, στους οποίους ε, οι γυναίκες εν γέννη και οι γυναίκες μετανάστριες πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαν να τύχουν περισσότερης προστασίας ε, και αναγνώριση της αξιοπρέπειά της. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο λοιπόν για το έργο σας. Ελπίζω να μπορέσετε αυτό να το συμμεριστείτε και με άλλα υπουργεία αντίστοιχα σε άλλες χώρες, διότι πραγματικά τη χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουρμάη στη συνέχεια για δύο λεπτά, το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Είμαι πολύ ευτυχής που σας υποδεχόμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ. Νιώσατε την κακομεταχείριση στο ίδιο σας το σώμα. Ξέρετε λοιπόν γιατί θέμα αναφερόμαστε εδώ. Όντως υπάρχει θέμα αλληλεγγύης, υπάρχει δημοκρατική κρίση, περισσότερη μυσαλλοδοξία. Χρειάζεται λοιπόν μια αλλαγή νοοτροπίας, πολιτιστική νοοτροπία. Και βεβαίως υπάρχουν ε, αλλαγές ε, στη νέα γενιά. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι πραγματικά το σχολείο είναι ένας τόπος όπου πολλά μπορούν να γίνουν. Όταν κοιτάξει όμως κανείς την ανώτατη εκπαίδευση, διαπιστώνει ότι υπάρχουν όλο και λιγότεροι άντρες. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι και εδώ θα πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα και συμφωνώ και με τις ερωτήσεις που έκανε η προηγούμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταραμπέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτά που έχετε υποστεί. Είναι μεγάλη τιμή για σας, για την Ιταλία που σας διόρισε σε αυτή τη θέση. Εγώ είμαι Βέλγος, αλλά ε, η οικογένειά μου είναι Ιταλικής καταγωγής και βεβαίως συνδέομαι ιδιαίτερα με τη χώρα σας. Θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ παράξενο το ότι έχετε υποστεί αυτές τις επικρίσεις. Εσείς στην Ιταλία. Στην Ιταλία που πραγματικά είναι μια χώρα που έχει γνωρίσει τεράστια κύματα μετανάστευσης πάνω από το μισό του πληθυσμού έχει αναγκαστεί κάποια στιγμή να μεταναστεύσει. Ενώ υπάρχουν 60 εκατομμύρια Ιταλοί αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Αναφερθήκατε σε κάποιες ε, νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσατε για την συμβασή της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει κυρωθεί τον Ιούνιο από ό,τι ξέρω. Μιλήσατε επίσης για οδηγίες, μιλήσατε για την ισότητα αποδοχών. Και σήμερα βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ενώ η συνθήκη της δρόμης ήδη ορίζει την ισότητα άνδρων και γυναικών, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι στην πραγματικότητα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στη λιτότητα, σε μείωση των δημόσιων επενδύσεων. Μήπως θα έπρεπε πέρα της νομοθεσίας να ξεκινήσουμε μία πολιτική δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη, κάτι το καθοριστικό για την ενσωμάτωση κάποιων ομάδων. Μήπως αυτός είναι ο τρόπος έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε σχέση και με τους νόμους που ψηφίζονται. Πρόεδρος, θα σας δώσω το λόγο, μπορείτε να απαντήσετε στα σχόλια και στις ερωτήσεις που ακούσαμε. Ναι. Η πρώτη ερώτηση για την κύρωση της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης. Η κύρωση έγινε στις 19 Ιουνίου. Η Ιταλία ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό και με το θέμα της βίας κατά των γυναικών, προσπαθώντας ε, ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία ε, έχει και θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της. Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες, ε, για το Υπουργείο το δικό μου, οι πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναλυφθούν ώστε οι γυναίκες μετανάστριες οι οποίες σε αυτή τη στιγμή είναι οι πιο ευάλωτες και αυτές που δεν ε, διαθέτουν ίσως την κατάλληλη κατάρτιση στοχεύουμε ιδιαίτερα και στην εκμάθηση της γλώσσας, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για την ένταξή τους σε οποιαδήποτε διαδικασία ενσωμάτωσης, είτε ε, από εργασιακής πλευράς είτε από κοινωνικής πλευράς. Ε, Σφέρεται λοιπόν ε, εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους δήμους και σε όλες τις περιοχές. Δυνατότητα κύκλων μαθημάτων που μπορούν να διατίθεται στις γυναίκες αυτές ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιφέρειες ε, και ε, περιοχές ε, συμμετείχα σε συναντήσεις επιχειρήσεων που στόχο έχουν την επιμόρφωση των γυναικών και κυρίως των γυναικών μεταναστριών διότι υπάρχει αυτή η ανισότητα παρά το γεγονός ότι υπάρχει ε, αρκετό υλικό από πλευράς νομοθεσίας, αλλά ε, είναι λυπής η εφαρμογή. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την ε, εκπαίδευση και την επιμόρφωση των γυναικών. Όσον αφορά την εμπορία των γυναικών. Υπάρχει πολύ προηγμένη νομοθεσία από πλευράς Ιταλία για την εμπορία γυναικών. Όσον αφορά τις γυναίκες μετανάστρες, ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα επόμενο βήμα. Δηλαδή να θεωρήσουμε πολλές γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε κέντρα κράτηση και κέντρα απέλασης, οι οποίες ορισμένες φορές βρίσκονται λανθασμένα σε αυτά τα κέντρα, διότι δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ε, είναι αδύναμες. Ε, πρέπει κάπως να διαφύγουν από αυτή την αγορά της εμπορίας ε, και επειδή είναι παράνομα στη χώρα, εμείς τις κλείνουμε στα κέντρα κράτησης και τις αποδυναμώνουμε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτούν καταλήλως και να προσπαθήσουμε να τις βοηθήσουμε να ενσωματωθούν ε, και πέραν από το θέμα της παρανομίας να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε να ξεφύγουν από τη δουλεία την οποία βιώνουν, διότι είναι πολύ προηγμένη νομοθεσία στην Ιταλία στο θέμα αυτό και προστατεύει τις γυναίκες. Όσον αφορά το διαφυλατικό διάλογο, ε, το Υπουργείο μου εδώ και μία εβδομάδα ασχολείται και με τις ε, πολιτικές για τους νέους πέραν των πολιτικών ε, ένταξης. Επομένως, θα είναι μια διπλή πρόκληση να ασχοληθώ για τις πολιτικές για τους νέους και για την ενσωμάτωση, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το διαφυλετικό διάλογο μέσω στήριξης και των πολιτικών για τους νέους για να μπορέσουμε να εντάξουμε και τους νέους στην αγορά εργασίας. Και η κυβέρνησή μας κάνει πάρα πολλά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, ε, συνεργάζεται και με το Υπουργείο Εργασίας, επενδύει πολλά στους νέους, πολλά στην εργασία των νέων και το Υπουργείο μου θα μπορέσει να κάνει και πάρα πολλά ε, για την ε, πολιτιστική αλλαγή, επενδύοντας τις κατάλληλες πολιτικές για τους νέους. Ένα τελευταίο στοιχείο, μια τελευταία ε, παρατήρηση με την οποία συμφωνώ απόλυτα, το γεγονός ότι η Ιταλία ήταν πάντα χώρα μετανάστευσης και σήμερα είναι μια χώρα που βιώνει τη μετανάστευση από την αντίστροφη πλευρά και αυτό λήφθηκε δεόντως υπόψη από τον Πρωθυπουργό Λέτα, διότι και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω διότι ήταν μακρόπνο το όραμά του και αντιλήφθηκε ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην Ιταλία έδωσε το μήνυμα και εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει μετανάστευση. Εγώ γεννήθηκα σε μια άλλη ήπειρο, κατάγομαι από άλλη χώρα αλλά σήμερα είναι Ιταλίδα. Πρόκειται λοιπόν για ένα παράδειγμα ενσωμάτωσης το οποίο θα πρέπει ε, να προβληθεί σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως αφορά και όλους τους μετανάστες που έχουμε εμεί στο εξωτερικό. Εγώ θεωρώ ότι μέσω του διορισμού μου, μέσω της κατάστασης της μετανάστευσης στην Ιταλία πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε έναν ολοένα και πιο στενό διάλογο και με πολλούς από τους Ιταλούς ε, που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν ε, μια πολύ προχωρημένη διασπορά και θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε επαφές και με άλλες χώρες ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά και να καταπολεμήσουμε και το ρατσισμό, μιλώντας με τους Ιταλούς μας στο εξωτερικό που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν τα μάλα, διότι πραγματικά μπορούν να αποδείξουν τι σημαίνει να φύγει κάποιος από τη χώρα του και να επιλέξει μια άλλη γη. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσει να συνεισφέρει σε αυτό και η Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ και εγώ που ήρθατε σήμερα εδώ σε εμά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μα και εμπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σα, σε όσους τομεί ε, γίνεται και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ε, ιδιότητα του Υπουργού. Okay, dear, uh, members. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής, θα αρχίσουμε τώρα την ψηφοφορία. Έχουμε δύο διαφορετικές ψηφοφορίες. Καταρχάς να πω ότι το σημείο 7 πρέπει να αναβληθεί για μετά την ψηφοφορία. Αρχίζουμε λοιπόν με το σημείο 8 της ημερησίας διάταξης για ισότητα ευκαιριών και ισότητα μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας. Κυρία Μπάουερ, ως εισηγήτρια θα θέλατε να πάρετε το λόγο ή να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ναι, προς επεξήγηση μόνο. Βλέπω και την κυρία Ζούμπερ εδώ. Να πω ότι εμείς ζητήσαμε ψηφοφορία κατά τμήματα για τις ε, συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα. Ζητήσαμε την ψηφοφορία κατά τμήματα για να καταλάβουμε στην ουσία τι συμβαίνει και ο λόγος είναι ότι στην μελέτη προσθεθέμενης αξίας που πήραμε Φάνηκε ξεκάθαρα ότι το ζήτημα των, του μισθολογικού χάσματος είναι πολύ σημαντικό, όμως ε, δεν ασχολούμαστε αρκετά με αυτό. Εάν λοιπόν ψηφίσουμε και συμπεριλάβουμε τις ε, συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις, δεν θα έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα όσον αφορά την προσπαθή για μείωση του μισθολογικού χάσματος. Ευχαριστώ πολύ. Α αρχίσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12, προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική αυτή τροπολογία. Όχι, ας την ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις για να προχωρήσουμε. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Είναι ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 3. Δεύτερο τμήμα. το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα όλο το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιανακουδάκη. Δεν σας άκουσα. Sorry, my car... Ναι, η κάρτα μου δεν λειτουργεί. Δεν έχει σημασία όμως, έτσι κι αλλιώς θα ψήφισα κατά. Υπολογίστε το λοιπόν. Θέλετε να το σημειώσουμε, ναι. Θα το σημειώσουμε και θα σημειώσουμε και την ψήφο υπέρ της κυρίας Κορνέλισεν. Επόμενη ψηφοφορία, σημείο 9 της μερίσιας διάταξης για τον εθελοντισμό και εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Αρχίζουμε με την τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51, υπέρ, κατά, αποχές, Ναι, ξέρω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Σε... Μπλοκ τροπολογία 51, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης ενημέρωση από την Επιτροπή Γυναικών σχετικά με την επίσκεψη στην Πορτογαλία. Okay, uh, Υπάρχουν πολλά μέλη που θέλουν το λόγο. Έχω τον κατάλογο εδώ. Αρχίζουμε με την κυρία Γκούρμα, η οποία ήταν ένα μέλο τη αντιπροσωπεία στην Πορτογαλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Πυκνό θα έλεγα. Και μετά από αυτό ετοιμάσαμε ένα πολύ καλό ενημερωτικό φυλάδιο για την κατάσταση. Φυσικά οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, λόγω της εμή προοδευτικής αγοράς εργασίας, βρίσκονται σε... Παρακαλώ, ησυχία. Δεν ακούω. Πρόεδρος, ε, κυρία Γκορμά έχει δίκιο. Παρακαλώ, ησυχία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σεβασμός. Όταν δεν ακούω τη φωνή μου υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, με χαρά μου ήμουν μέλο τη αντιπροσωπεία. Το πρόγραμμά μα ήταν αρκετά πλούσιο. Οι συνάδελφοι ήταν εξαιρετικοί. Φυσικά είχαμε και την αντιπρόεδρο, την Edit, η οποία σύνταξε ένα πολύ επαγγελματικό πρόγραμμα. Με ανησυχία, όμω πάρα πολύ η κατάσταση στην Πορτογαλία για την κρίση. Ήδη συζητήσαμε και αναφέραμε ότι αυτή η κρίση είναι υφέρπουσα και επηρεάζει τις γυναίκες περισσότερο. Ελπίζω όμως να έχουμε και στο μέλλον εξίσου καλές αντιπροσωπείες και εξίσου καλά επαγγελματικά προγράμματα και να επιστρέψουμε. Ας ελπίσουμε λοιπόν να υπάρχει μια αλλαγή της κυβέρνησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Κυρία Στρέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την κυρία Γκορμάη, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικά δραστήρια και ήμασταν σε επαφή με μέλη ενώσεων, οργανώσεων, και ενώσεις ε, που προστατεύουν και προσφέρουν βοήθεια στα θύματα κακοποίησεων και βίας. Επίσης ήρθαμε σε επαφή και με την πλατφόρμα των γυναικών. Ήρθαμε σε επαφή με την ε, Κυβερνητική Επιτροπή για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και συναντηθήκαμε με την πρόεδρο του αρμόδιου οργανισμού για την ε, παρακολούθηση αν θέλετε, μια ομάδα που ανήκει στην επιθεώρηση εργασίας, παρακολούθηση για, την, για το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που πλήττει κυρίως τις γυναίκες, αυτό που είδαμε στην Πορτογαλία είναι ότι όντως οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευάλωτες και εκτίθενται περισσότερο στις διακρίσεις. Και ότι υποφέρουν περισσότερο από την αλλεργία, ότι δυσκολεύονται με την ανατροφή των παιδιών και πραγματικά συγκινηθήκαμε ιδιαίτερα με κάποιες πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις που είδαμε. Υπάρχουν γυναίκες, παραδείγματο χάρη, που προσπαθούν να ενσωματωθούν ε, στην αγορά εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα και δεν ε, μπορούν να υποφεληθούν από στοιχειώδη δικαιώματα, όπως παραδείγματο χάρη η ε, αδιαμητρότητας. Και φυσικά και αναφέραμε τις περιπτώσεις αυτές, τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες μας διασφάλισαν και μας επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν έλεγχοι και ότι φυσικά τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εντοπίζονται και να υπάρχουν κυρώσεις. Επίσης μιλήσαμε και με την υφυπουργό, τον υφυπουργό συγγνώμη, αρμόδιο για τις γυναίκες και την απασχόληση για τις περιπτώσεις ε, γυναικών που δεν έχουν απολύτως κανένα επίδομα το τοκετού είτε μπορούν να απολυθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους χωρίς απολύτως καμία αποζημίωση. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης ήταν πολύ ε, χρήσιμα, πολύ επικοδομητικά και φυσικά και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ε, ενώσεις αυτές που συναντήσαμε έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις γυναίκες από τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα αυτής της κρίσης έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση των γυναικών και να μην επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η οικονομική τους κατάσταση στην Πορτογαλία. Δυστυχώς το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Πορτογαλίας βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και ο μεγαλύτερος αριθμός αυτού του πληθυσμού είναι γυναίκες. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι η επιδείνωση της κατάστασης των γυναικών έχει επιπτώσεις και στα παιδιά. Πολλά παιδιά σήμερα τρώνε μία φορά την ημέρα ζεστό μαγειρεμένο φαγητό και αυτό είναι το μεσημέρι στο σχολείο. Επίσης, βλέπουμε πολλά παιδιά τα οποία καταφεύγουν στο σχολείο γιατί δεν μπορεί η οικογένειά τους να τα προστατεύσει και να τους παρέχει τα στοιχειώδη. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να παρακολουθήσουμε προσεκτικά την κατάσταση έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε με το σημείο 7 που αφορά την αντιπροσωπεία στην Πορτογαλία, η κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι που συμμετείχαν και αυτές στην αντιπροσωπεία. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω κάποια σημεία και να μετριάσω λίγο την αποσιοδοξία που εκφράστηκε υπήρξε όντως η επίσκεψη της αντιπροσωπείας, ε, πολύ σημαντική επίσκεψη και για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη ε, ποιες είναι οι συνέπειες της κρίσης στην ισότητα των φίλων και στις ίσες ευκαιρίες στην Πορτογαλία. Πρόκειται για μια επίσκεψη η οποία εστίασε σε συγκεκριμένα θέματα και πέραν των όσων ακούσαμε από τις συναδέλφους, οι οποίες ε, μίλησαν προηγουμένως, έγινε και μια πολύ σημαντική συνάντηση με την Τερέζα Μωράης, υπεύθυνη για κοινοβουλευτικά θέματα και ίσες ευκαιρίες. η οποία μας έδωσε κάποια παραδείγματα για την κατάσταση των γυναικών. Έκανε μία αντιπαράθεση μεταξύ της κατάστασης των γυναικών προ-κρίσης και μετά-κρίσης και είπε ποια είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η πορτογαλική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες ε, φυσικές δυσκολίες από τις οποίες πάσχει η πορτογαλική κοινωνία και πιο συγκεκριμένα οι γυναίκες στην Πορτογαλία. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει το μνημόνιο της Τρόικας, ε, το οποίο είναι σε διαδικασία εφαρμογής και αυτό φυσικά έχει και κάποιες συνέπειες. Διότι υπάρχει και υποχρέωση εξοικονόμησης χρημάτων. Η Γενική Γραμματέας μας είπε ότι υπάρχουν ε, καταστάσεις απόλυτης ένδυας, ε, οι οποίες ελοχεύει ο κίνδυνος να επιδεινωθούν λόγω της κρίσης και κυρίως όσον αφορά τις γυναίκες και πολλό δε μάλλον γυναίκες οι οποίες ε, ε, δεν έχουν μια θέση εργασίας, δυσκολεύονται να βρουν θέση εργασίας και ζουν μόνος. Ε, υπάρχει λοιπόν αύξηση της φτώχειας μεταξύ των γυναικών και η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι της τάξης του 12%. Ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 16%. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Όσον αφορά την πολιτική εκπροσώπηση, ε, υπήρξαν οι λεγόμενες ροζ ποσοστώσεις, ε, που σημαίνει ε, ότι είχαμε σημαντικά αποτελέσματα, διότι πριν τη συγκεκριμένη νομοθεσία μόνο 5% των βουλευτών ήταν γυναίκες, ενώ τώρα είναι πολύ πιο πολλοί άριθμες. Εκφράστηκε όμως και μία ανησυχία για την αύξηση των περιστατικών βίας ε, σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση λαμβάνει κάποια προληπτικά μέτρα μαζί και με τις αστυνομικές δυνάμεις ε, προκειμένου να προβλέψει αυτή την ε, χαρακτηριστική αύξηση που παρατηρείται σε ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, κατά γυναικών όταν δηλαδή υπάρχει κοινωνική και οικονομική κρίση. Συναντηθήκαμε επίση και με κάποιε οργανώσει οι οποίε μα έδωσαν μια πολύ αντικειμενική εικόνα του τι ακριβώ συμβαίνει στην Πορτογαλία. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να πω ότι η Πορτογαλία προφανώ και βρίσκεται σε μια κατάσταση κρίση. Αυτό δεν ωφελεί κανέναν και σίγουρα δεν ωφελεί τις γυναίκες. Αλλά οι εθνικές αρχές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για τις γυναίκες ε, στην Πορτογαλία. Η κυρία Τζούμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να συμφωνήσω κι εγώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Πορτογαλία. Και αυτό ε, φάνηκε και το αντιλήφθηκαν όλοι όσοι συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία μπορέσαμε να κάνουμε μία διάγνωση της κατάστασης των γυναικών στην Πορτογαλία και πέραν των ε, συνεδριάσεων με θεσμικούς φορείς, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση με τις οργανώσεις οι οποίες εργάζονται επί τόπου, πολύ συχνά σε δύσκολες συνθήκες, οι οργανώσεις αυτές ε, γνωρίζουν πράγματα τα οποία δεν προβάλλονται τόσο καλά στα στατιστικά στοιχεία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που τάραξε περισσότερο και εντυπωσίασε περισσότερο τις συναδέλφους, οι οποίες δεν κατάγονταν από την ε, Πορτογαλία, ήταν το γεγονός ότι στη διάρκεια των συναντήσεων οι γυναίκες μας είπαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με τις συνέπειες της κρίσης, αλλά και με τις συνέπειες ε, των στρατηγικών και των μέτρων τα οποία έλαβε η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες και τελικώς πολλές φορές καταλήγουν να οξύνουν τα προβλήματα. Ε, υπάρχουν προβλήματα σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε δημόσιες υπηρεσίες, ελήφθησαν κάποια μέτρα τα οποία ε, μειώνουν τους μισθούς, ε, δεν υπάρχει αρκετή κοινωνική βοήθεια, μειώθηκαν κάποια επιδόματα και επομένως ε, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόζει κάποιος τέτοια μέτρα και στη συνέχεια να λέει ότι α, ανησυχούμε γιατί υπάρχει ανισότητα για μεταξύ της μισθολογικής κατάστασης ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν επίσης γυναίκες οι οποίες είναι θύμα οικογενειακής βίας και βρίσκονται στο σπίτι του ανθρώπου που τους επιτίθεται, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν οικονομική ανεξαρτησία, πολύ λιγότερο δε σε σχέση με το παρελθόν. Η προοπτική λοιπόν μιας αυτονομίας για τις γυναίκες είναι πολύ μικρότερη πλέον. Είναι υποχρεωμένες λοιπόν να συμβιούν στο ίδιο σπίτι με τον άνθρωπο ο οποίος ε, τις κακομεταχειρίζεται. Υπήρξαν αρκετές μαρτυρίες και μας έκαναν έναν απολογισμό οργανώσεις ε, ε, οι οποίες ασχολούνται με γυναίκες που βρίσκονται σε αυτές τις ε, συνθήκες. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες εξωθούνται στην πορνεία λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να θρέψουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να ζητούμε από κανέναν να κάνει τέτοιες θυσίες. Ευχαριστώ κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ βρήκα εξαιρετικά χρήσιμη και σημαντική την αποστολή μας στην Πορτογαλία. Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό, ήταν ε, πολύ επίπεδο και μας έδωσε μια πολύ καλή εικόνα της κατάστασης στην Πορτογαλία. Να σας υπενθυμίσω ότι η Πορτογαλία έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση και η νεολαία πολλές φορές αναγκάζεται να γυρίσει στο σπίτι των γονιών ή ακόμα και των παππούδων τους και αναλογιστείτε τι σημαίνει να ταΐζεις μια οικογένεια με μια πολύ πολύ μικρή σύνταξη επειδή τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου δεν έχουν δουλειά εξαιτίας της κρίσης. Τότε πιστεύω πως έχοντας αυτό υπόψη θα δοθεί η δυνατότητα να μας ανοίξουν τα μάτια γιατί πραγματικά υπάρχει διαπραγματευτική ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βέρτμαν. Μπορούμε να προχωρήσουμε, πιστεύω, και να περάσουμε στο σημείο 11 προτείνω, προτού ασχοληθούμε με το σημείο 10. Θα εξετάσουμε λοιπόν την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών πρώτα και έπειτα την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγραμματός της Στοκχόλμης. Αν το δέχεστε τότε πάμε κατευθείαν στο σημείο 11, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Και αυτό που θα ήθελα τώρα είναι να δώσω το λόγο στη νομική υπηρεσία στον Αντώνιο Κάουλα, επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την νομική μας εκνομοδότηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, συναδελφό μου τον Πασκάλ Σονάρ που ε, με βοήθησε στην νομική γνωμοδότηση και τη συνταξή της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που έχουμε να παρουσιάσουμε την νομική μας γνωμοδότηση για την νομική βάση μιας πρωτοβουλίας καταπολέμησης της βία κατά των γυναικών σε απλής ποινικού δικαίου. δικαίου. Συμπεράναμε ότι στις ε, συνθήκες δεν υπάρχει κάποια γενική νομική βάση για νομοθετική πράξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση βίας ε, προς ε, τι γυναίκε από πλευρά ποινικού δικαίου. Ωστόσο, Βρήκαμε επίσης ότι σε ορισμένους τομείς πολιτικής ενδεχομένως να υπάρχει βάση για κοινοτική νομοθεσία ποινικού δικαίου που να σχετίζεται με την καταπολέμηση βίας κατά των γυναικών, μόνο όμως σε ορισμένα, μόνο όμως σε βία που γίνεται σε ορισμένο ε, πλαίσιο. Δηλαδή, σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών συμπεριλαμβανόμενης της ε, βίας που σχετίζεται με την ε, προετοιμασία, διευκόλυνση, συνοδεία και κάλυψη σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, περιοχές οι οποίες είναι ήδη αντικείμενο ε, νομοθεσίας κατά των διακρίσεων φύλου, δηλαδή στους τομείς της απασχόλησης, ε, της επαροχής αγαθών και υπηρεσιών και τέλος υποστηρικτικά μέτρα για την πρόληψη του εγκλήματο. σε τομεί όπου τα κράτη-μέλη ήδη είναι ενεργά στην καταπολέμηση τη βίας ε, προς τις γυναίκες. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου τώρα να συνοψίσω το σκεπτικό πίσω από το οποίο ε, έχουμε οδηγηθεί σε αυτά τα συμπεράσματα. Σύμφωνα με την ε, αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 της συνθήκης, κάθε νομική πράξη προς έγκριση από το νομοθετικό σώμα της Ένωσης απαιτεί να υπάρχει νομική βάση. Μόνο διατάξεις των συνθήκων που δίνουν ε, συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο νομοθετικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να υπηρετήσουν ως νομική βάση. Αυτό αποκλεί ευθύ εξ αρχή σε διατάξεις οι οποίες αναφέρονται σε στόχους και αξίες όσο και αναγκαίο να είναι να υπάρχει κάποια καθοδηγητική γραμμή για την Ένωση. Παρομοίω, τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, παρότι είναι δεσμευτικά ε, για την Ένωση, όποτε η Ένωση έχει το δικαίωμα να δράσει, δεν δίνουν το δικαίωμα αυτά καθ' αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει. Αυτό ευκρινίζεται στο, στις διατάξεις του άρθρου 51, παράγραφος 2 της χάρτας, θα σας το διαβάσω, λέει... Λοιπόν, ότι η χάρτα δεν επεκτείνει το ε, το, το πεδίο εφαρμογή κοινοτική νομοθεσία πέρα από τι ε, εξουσίε τη Ένωση ούτε δημιουργεί νέο ε, όργανο ή νέο όργανο για την Ένωση, ούτε τροποποιεί αρμοδιότητες και εξουσίες όπως αυτές ορίζονται από τις συνθήκες. Έτσι λοιπόν, εκτός από την χάρτα, έπρεπε να αναλύσουμε και πολιτικές, τομεακές πολιτικές, όπως για παράδειγμα το άρθρο 19 της συνθήκης, Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των διακρίσεων. Μια διάταξη που γνωρίζετε πολύ καλά εσείς στην Επιτροπή σα. το άρθρο 153 παράγραφο 2 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Αυτά θα μπορούσαν να είναι κάτι ενδιαφέρον για να δημιουργηθεί νομική βάση, όμως το συγκεκριμένο ζήτημα του ποινικού δικαίου δεν μας βοηθούν ούτε αυτά, διότι υπάρχουν πιο συγκεκριμένε διατάξει ποινικού δικαίου στην συνθήκη σε άλλα σημεία. Η συνθήκη τώρα προβλέπει ένα κεφάλαιο για δικαστική συνεργασία σε θέματα ποινικού δικαίου, το οποίο έχει άλλων νομικών βάσεων όσον αφορά τους ορισμούς των αξιοπινών πράξεων, τις ποινικέ κυρώσει και συγκεκριμένα μέτρα πρόληψη του εγκλήματο. Έτσι λοιπόν, μόνο αυτέ οι νομικέ συμβάσει του τελευταίου κεφαλαίου για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικά ζητήματα μπορούν ενδεχομένω να είναι χρήσιμα για αυτό που εσά ενδιαφέρει. Και η συγκεκριμένη νομική βάση την οποία σκεφτόμαστε είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 83, η παράγραφο 2 του άρθρου 83 και το άρθρο 84 τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα, τις θα αναλύσω αυτά τα άρθρα από την αρχή. Αρχίζουμε με το άρθρο 84. Αυτή... Αυτό είναι νομική βάση για συμπληρωματικά μέτρα για την πρόληψη του εγκλήματος, δηλαδή να υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη μόνο σε δράσεις. Θα μπορούσε να είναι μια κατάλληλη νομική βάση για μια νομοθετική πράξη που θα παρέχει κανόνες ανταλλαγής και συλλογής πληροφοριών, κατάρτισης των ε, αρμόδιων αρχών, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, ευαισθητοποίησης, ε, δημιουργίας ταμείων κτλ. Σε σημείο που αυτές μπορούν να ε, προωθούν ή να στηρίξουν τις δράσει των κρατών μελών για την ε, πρόληψη εγκλημάτων βίας κατά των γυναικών. Ωστόσο, να είμαι σαφή, το άρθρο 84 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλεί οποιαδήποτε εναρμόνιση νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν ιδιαίτερα το άρθρο 84 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει ε, ποινικά δικήματα ή να ε, αναφέρεται σε κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, άρθρο 83 παράγραφος 1. Εδώ έχουμε μία διάταξη η οποία θα μπορούσε ενδεχομένω να μας επιτρέψει να ε, υιοθετήσουμε ελάχιστου κανόνε για τους ορισμούς και τις κυρώσει ποινικών αδικημάτων, όμω μόνο σε ορισμένου, συγκεκριμένου, ρητά ε, αναφερόμενους για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα. Το άρθρο 83 παράγραφος 1 δεν αναφέρει βία που σχετίζεται με το φύλλο ή βία κατά των γυναικών ως εγκλήματα τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν τέτοια νομοθεσία. Έτσι, και το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ε, Σύνθηκης Λειτουργίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για γενικές ε, ε, διατάξεις ποινικού δικαίου για τη βία κατά των γυναικών, εκτός αν το Συμβούλιο ομόφωνα προσέθεται ένα τέτοιο έγκλημα στην, στον κατάλογο. Ωστόσο, το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται σε εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών και, σε, και στο οργανωμένο έγκλημα. Έτσι, η βία κατά των γυναικών στο πλαίσιο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενδεχομένως μπορεί να υπόκειται σε ελάχιστους κανόνες ποινικού δικαίου όπως για βία κατά την προετοιμασία, διευκόλυνση ή κάλυψη σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε γυναικών. Το ίδιο ισχύει και για κανόνες ποινικού δικαίου για τη βία κατά των γυναικών στο συγκεκριμένο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος. Εδώ λοιπόν υπάρχει μία δυνατότητα που μας ε, δίδεται από συγκεκριμένο πλαίσιο. Τώρα, άρθρο 83, παράγραφος 2 της Συνθήκης Λειτουργίας. Εδώ Μα παρέχεται άλλη μια νομική βάση για τους κανόνες σε ορισμούς και κυρώσει ποινικού δικαίου, μόνο όμως σε συγκεκριμένους τομείς. Τομείς αυτοί εδώ είναι ε, ε, μέτρα εναρμόνισης και όπου το ποινικό δίκαιο ε, καθιστά αναγκαία τέτοια μέτρα εναρμόνισης, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικά. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν υπήρχαν ορισμένες εναρμονισμένες ε, πολιτικές και τομίσεις στο κοινοτικό δίκαιο, την αποτελεσματικότητα των οποίων θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε με ε, ποινικέ διατάξεις για τη βία κατά των γυναικών. Αυτό που βρήκαμε φυσικά μετά από λεπτομερή ανάλυση είναι ότι εδώ θα μπορούσε να ισχύει αυτό στις, ε, στους τομείς της απασχόλησης, και στον τομέα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Τώρα, όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία, η Οδηγία 2006-54, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά, θέτει μη ποινικού σε ε, συμπεριλαμβανομένε μιας απαγόρευσης διακρίσεων βασισμένη στο φύλλο, ε, στην απασχόληση και συνθήκες εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της παρενόχλησης, η οποία επίσης αναφέρεται σε αυτό το πλαίσιο και απαγορεύεται. Στη γνωμοδότησή μας λοιπόν επιχειρηματολογούμε και λέμε ότι η βία κατά των ε, γυναικών, εάν ασκείται ακριβώς επειδή το άτομο είναι γυναίκα, μπορεί να θεωρηθεί μία ιδιαίτερα ακραία μορφή διάκρισης. Γι' αυτό ενδεχομένως αυτή η οδηγία 2006 54 θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αναφέρεται ρητά για την βία κατά των γυναικών στον χώρο εργασίας. Επομένως, ως ε, συνέπεια αυτού, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι στο χώρο εργασίας λαμβάνει χώρα βία κατά των γυναικών παρά την οδηγία αυτή, υπάρχουν, υπάρχει ποινικό δίκαιο, υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες για αυτούς ε, τους ε, για αυτές τις περιπτώσεις οι οποίοι είναι ενδεχομένως να, ε, οι οποίοι είναι δυνατόν να, να χρησιμοποιηθούν κατά από το άρθρο 83 παράγραφος 2. Τώρα όσον αφορά την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Η οδηγία του 2004 113 περιλαμβάνει παρόμοια απαγόρευση των διακρίσεων βασισμένη στο φύλλο ως την οδηγία και την απασχόληση που ανέφερα πιο πριν. Αυτή η οδηγία 113 του 2004 περιλαμβάνει παρόμοιους ορισμούς για τις άμεσες διακρίσεις και για την παρενόχληση ως μία μορφή διάκρισης. Και εδώ λοιπόν, στον τομέα παροχής αγαθών και υπηρεσιών, πάλι ε, μόνο μετά από λεπτομερή ανάλυση, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 83 παράγραφος 2 ως νομική βάση για την, τον κλάδο παροχής αγαθών και υπηρεσιών και να μπορέσουμε έτσι να ρυθμίσουμε και την βία κατά των γυναικών. Τώρα θα ήθελα να συνοψίσω τα ευρήματά μας. Σύμφωνα με την νομική μας εγνωμοδότηση, δεν υπάρχει νομική βάση στις συνθήκες για ένα οριζόντιο ε, μέσω ποινικού δικαίου για την βία κατά των γυναικών. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπάρχει νομική βάση ή βάσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στο ποινικό δίκαιο στα πλαίσια σεξουαλικής εκμετάλλευσης, οργανωμένου εγκλήματος, απασχόλησης και παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Τώρα να προσθέσω κάτι Χρειάζεται προσοχή, διότι η ανάλυση μας αναφέρεται μόνο στο πεδίο εφαρμογή και των νομικών βάσεων που αναφέρθηκαν. Δεν αναλύσαμε τις υπόλοιπες ε, συνθήκες εφαρμογής, οι οποίες φυσικά θα πρέπει να συμμορφώνονται Ιδιαίτερα το άρθρο για την αποτελεσματικότητα, την παράγραφο 2 του άρθρου 83 και οι αναφορές στην επικουρικότητα και την αναλογικότητα σύμφωνα με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν στα πλαίσια του κειμένου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Thank you very much for... πολύ για την παρουσία αυτής της νομικής γνωμοδότησης. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Επιτροπή μας, γιατί για πρώτη φορά η νομική υπηρεσία κάνει μια τέτοια παρουσίαση νομικής ε, γνωμοδότησης. Μπράβο λοιπόν. Εντυπωσιαστήκαμε. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, σχόλια. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν τη νομική υπηρεσία που παρουσίασαν αυτή τη γνωμοδότηση. Ξέραμε από την αρχή ότι το θέμα δεν είναι απλό, είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Κάθε φορά που ζητήσαμε από την Επιτροπή και ήρθαμε σε επαφή και με την Επίτροπο, την κυρία Ρέντινγκ, οι δυσκολίες ήταν προφανείς και εκφράστηκαν και από την νομική υπηρεσία της ε, Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο παρόλα αυτά και η Επιτροπή μας, όλο το Κοινοβούλιο όμως επιμένω, έχει δεσμευθεί για την πρόθεση του θέματος αυτού. Και φυσικά και θα συνεχίσουμε στην προσπάθειά μας για να υπάρξει νομική βάση και να προωθηθεί το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Είναι ένα θέμα που είναι παρόν σε όλες τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν συζητούμε για θέματα ισότητας των φύλων. Απογοητεύομαι λοιπόν με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Ναι, εντάξει, ε, ε, επεξεργαστήκατε το θέμα, αλλά περιμέναμε κάτι παραπάνω. Και το ίδιο και όλα τα μέλη της Επιτροπής θα σας πούν. Στο Συμβούλιο σίγουρα θα υπάρξουν αντιρρήσεις. Εσείς όμως είστε η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και η δουλειά σας είναι να μας στηρίξετε. Εμείς λοιπόν θέλουμε να προωθήσουμε το θέμα και εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι και άλλες παρόμοιες εμπειρίες υπάρχουν εδώ. Η νομική υπηρεσία μπορεί να κάνει τα πάντα. Αναφερθήκατε στο άρθρο 83 και το 84. Όντως, αυτό που είπατε είναι σωστό, αλλά εμείς δεν περιμένουμε η σεξουαλική εκμετάλλευση, το οργανωμένο έγκλημα, η απασχόληση, η κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών να είναι ο κύριος τομέας όταν μιλάμε για ισότητα των φυλών. Ναι, έχετε δίκιο. Και αυτοί οι τομείς ε, μπορεί να αναφερθούν όταν μιλούμε για την ε, βία κατά των γυναικών. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τομέας όταν ε, πρόκειται για την ενδοοικογενειακή βία είναι κάτι διαφορετικό από το οργανωμένο έγκλημα, από την σεξουαλική εκμετάλλευση, από το χώρο εργασίας, όπου και εκεί μπορεί να υπάρχει αυτή η, αυτό το φαινόμενο. Προφανώς η κυκλοφορία, η διανομή αγαθών και υπηρεσιών, η ε, απασχόληση όντως να έχουν σαν συνέπεια την βία στο εσωτερικό μιας οικογένειας. Όλο και περισσότερες ενδείξεις μας οδηγούν στη διαπίστωση και περιμένουμε εξάλλου και από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μια έκθεση για τη βία. Τα στοιχεία πάντως είναι ανησυχητικά. Η κατάσταση είναι σοφερή και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανεξάρτητες μελέτες και έρευνες. Υπάρχει μια μελέτη που προετοιμάζεται εξάλλου νομική μένα, αλλά όχι από μια νομική υπηρεσία. Είναι μια έρευνα που βασίζεται στην εργασία κοινωνιολόγων. Εγώ πολύ θα ήθελα να δω τη δική τους νομική άποψη και γνωμοδότηση αλλά πραγματικά η Επιτροπή αυτή θέλει να εκφράσει την βούλησή της, την επιθυμία της, να δούμε ποιος είναι ο τρόπος να φτάσουμε σε μία νομική βάση, κοιτώντας άλλες οδηγίες και όχι μόνο αυτές τις δύο που μας αναφέρεται και οι οποίες καλύπτουν την απασχόληση και την κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. γιατί η σεξουαλική εκμετάλλευση δεν είναι, και το οργανωμένο έγκλημα, δεν είναι οι περιπτώσεις αυτές που μας απασχολούν περισσότερο και πιο συχνά όταν μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη γνωμοδότηση, αλλά περιμένουμε πολύ περισσότερα. Νομίζω μπορείτε να μας βοηθήσετε καλύτερα και να μας ε, ε, καθοδηγήσετε σε αυτό που περιμένουμε. Να κάνετε, εν πάση περιπτώσει, αυτό για το οποίο έχετε προσληφθεί, που είναι να εργαστείτε στην ε, υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να προσπίσετε τα αιτήματά μας. Πραγματικά είστε η συγκήτρια του θέματος αυτού, το αποδείξατε η κυρία Μπιλμπάου έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, βρισκόμαστε ενώπιον ενός ε, θέματος το οποίο είναι πολιτικά ορθό και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάθε εβδομάδα, κάθε φορά όλοι αναφερόμαστε στην ανάγκη να προχωρήσουμε και να καταπολεμήσουμε την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά όλες τις πληροφορίες της νομικής υπηρεσίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση που μας μοιράστηκε. Αυτοί έκαναν τη δουλειά τους, μπορούμε να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε λίγο πολύ. Εγώ όμως θα ήθελα να ρωτήσω το εξής αν όλες οι οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνουμε τους τελευταίους μήνες ε, συνεπία μιας ε, ακραίας κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμπίπτουν στην συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματο χάρη, χρηματοπιστωτική εποπτεία ή μέτρα τα οποία ε, λήφθησαν στη δέσμη των 6 μέτρων ή τη δέσμη των 2 μέτρων. Αν εξετάσουμε το καθένα ξεχωριστά, σίγουρα θα βρούμε μια αντίστοιχη η γνωμοδότηση ε, νομική από οικονομική σκοπιάς ε, με αυτήν που ακούσαμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Εδώ πρόκειται για πολιτική απόφαση. Όταν ε, πρόκειται για οικονομικά ζητήματα φαίνεται ότι είναι πολύ εύκολο να υπερβούμε τη συνθήκη λειτουργίας της Ένωσης και δεν θέτουμε ζητήματα τα οποία δυσκολεύουν την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όταν πρόκειται κυρίως για γυναίκες, γιατί εδώ πρωτίστως ε, το πρόβλημα είναι των γυναικών, ε, πάντα τα προσκόμματα είναι πολύ περισσότερα. Δεν έγινε και τίποτα βέβαια, γιατί συνηθισμένες είμαστε. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να πω ότι η βία κατά των γυναικών σε πολλές χώρες ήταν κάτι το οποίο χρειάστηκε να επεξεργαστούμε πάρα πολύ, διότι η βία ε, λόγω φύλου, την οποία συζητούμε τώρα, που δεν έχει καμία σχέση με την εκμετάλλευση των γυναικών, ούτε το οργανωμένο έγκλημα, ε, η βία στον ε, ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό χώρο ήταν κάτι το οποίο χρειάστηκε να επεξεργαστούν πολλές κυβερνήσεις ώστε να φτάσει πλέον και να συζητείται δημόσια σε κάθε κράτος μέλος αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι έχει φτάσει πλέον η στιγμή εντό τη Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την οποία δημιουργούμε και σε οικονομικό επίπεδο, να κάνουμε και αυτό το άλμα για την καταπολέμηση της ανισότητας κατά των διακρίσεων και κυρίως κατά το εισβίας λόγω φύλου. Και αυτό θα πρέπει να προβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε ότι τα στοιχεία τα οποία ανέφερε η κυρία Παρβάνοβα σε αυτές τις αιτήσεις εκθέσεις είναι πραγματικά σκανδαλώδη. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μαθαίνουμε νέα σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιφέρειες, σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά της Ευρώπης. Ξυπνάμε με ανακοινώσεις δολοφονιών γυναικών. Και εδώ δεν συμβαίνει τίποτα θεωρείται ως μη Αλλά αν γίνει μια απόπειρα ή οποιαδήποτε, τότε ξαφνικά είναι σκάνδαλο. Και συμφωνούμε γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Αλλά τα ποσοστά των γυναικών που δολοφολούνται ετησίω φαίνεται ότι δεν μας ενδιαφέρουν από πολιτική σκοπιά, διότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ασχοληθούμε με το ζήτημα. τούτου λεχθέντος και λαμβάνοντας υπόψη το θετικό στοιχείο το οποίο ανέφεραν ε, οι συνάδελφοι από την νομική υπηρεσία. Αναφέρθηκαν στα άρθρα τα οποία θα μπορούσαν ε, να μας απασχολήσουν και θα μπορούσαμε να εξετάσουμε από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέγεται ότι υπάρχει μια δυνατότητα που είναι το Συμβούλιο ομόφωνα να αποφασίσει να εγκρίνει το συγκεκριμένο θέμα. Και προσωπικά, επειδή θεωρώ ότι όλοι εδώ στην Επιτροπή μας είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να γίνει αυτό το άλμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών, η οποία πολύ συχνά συνοδεύεται ε, και με την ισότητα, θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορεί να μας συμβουλεύσει η νομική υπηρεσία ώστε εμείς από πλευράς Επιτροπής μας να προτείνουμε στο Συμβούλιο να ε, εντάξει ή να διευρύνει ε, ε, τον κατάλογο με τα στοιχεία που έχει. Και θα τους ήμασταν ευγνώμονες. Ευχαριστώ η κυρία Χιμένεθ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου του Κοινοβουλίου συγγνώμη, για την γνωμοδότηση. Ε, συνεργαστήκαμε στην ε, οδηγία για την ε, στήριξη και προστασία των θυμάτων σοβαρών εγκλημάτων και είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ μαζί τους και να δω πώς εργάζονται και εδώ πρέπει να πω ότι πρόσεξα και με αυτό συμφωνώ με την κυρία Παρβανόβα ότι αναφέρθηκε η βία κατά των γυναικών στην απασχόληση, στις υπηρεσίες, σαφώς και τη σεξουαλική εκμετάλλευση που είναι αναπόσπαστο τμήμα ε, των εγκλημάτων αυτών, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις βίας κατά γυναικών είναι οικογενειακή βία. Μπορεί να είναι ε, βία του ζεύγους, μπορεί να είναι από κάποιον από το φιλικό περιβάλλον, αλλά από ό,τι φαίνεται συνήθως συμβαίνει εντός της οικογένειας και των φιλικών σχέσεων. Εάν δεν ασχοληθούμε λοιπόν με αυτό το θέμα, θεωρώ ότι είναι χωρίς νόημα συγκεκριμένη οδηγία. Πρέπει να βρούμε λοιπόν κάτι ώστε να καλύψουμε και αυτή την, ψυχή, την πτυχή. Ε, εγώ βρήκα τα πράγματα εύκολα στην οδηγία με την οποία ασχολήθηκα υπήρχε πολύ μεγάλη στήριξη και εκεί υπήρχε και ένα κεφάλαιο που αφορούσε τη βία κατά των γυναικών και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το εντάξουμε και αυτό εκεί. Θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι θεωρούμε ότι πρέπει η βία κατά των γυναικών να θεωρηθεί έγκλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι το θέμα. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα επ' αυτού. Και θα ήθελα να ζητήσω πώς μπορούμε εμείς από το Κοινοβούλιο να κάνουμε μια απόπειρα να παρουσιάσουμε κάτι στο Συμβούλιο και θα το δεχτεί προς αυτή την κατάσταση, να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα. Ξέρω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ήταν σαφής η επιθυμία του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εγκλήματα τα οποία ε, πλήττουν την κοινωνία μας καθημερινά, ε, άλλες φορές μειώνονται, κάθε χρόνο μειώνονται λίγο, μετά ξανανεβαίνουν, εξαρτάται από ε, τις κυβερνήσεις. Ε, δεν μπορεί όμως κανείς ε, να αντιμετωπίσει από πολιτική σκοπιά στο ζήτημα. Και υπάρχει όμως και ένα πάγιο αίτημα από πλευράς κοινωνίας να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό. Εγώ θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια την κυρία Παρβανόβα για την έκθεση αυτή και θα συνεχίσουμε όλοι μαζί να ε, βοηθούμε για το θέμα αυτό. Η κυρία Αντζελίλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παρφανόβα για την αποφασιστικότητα ε, με την οποία προσπάθησε μαζί με τις υπόλοιπε συναδέλφους να προχωρήσει κάτι το οποίο πρέπει εξορισμού να είναι φιλόδοξο. Δεν ε, θέλουμε απλώς να φτιάξουμε μια ωραία έκθεση, αλλά θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι και Ακριβώς γι' αυτό βασιζόμαστε και στην υποστήριξη της νομικής υπηρεσίας, η οποία ήδη έχει κάνει αρκετά. Μας έδωσε κάποια ενάψματα, κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, με πάσα προσοχή βέβαια, αλλά έκανε πολλά και μας βοηθά. Θα θέλαμε όμως να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι όταν ε, ξεκίνησε η συγκεκριμένη θητεία, είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες ενώπιόν μας. Αλλά καταφέραμε να περάσει οδηγία για την εμπορία ανθρώπων, για την οδηγία των θυμάτων, το ένταλμα προστασίας, η οδηγία για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και την παιδοπορνογραφία. Όλα αυτά είναι πράγματα συγκεκριμένα τα οποία εκτιμούν οι πολίτες διότι αφο, τους αφορούν πολύ συγκεκριμένα. Ακόμα και όταν ξεκίνησε η συζήτηση για το τράφικινγκ και την εμπορία ανθρώπων υπήρχαν πολλά προβλήματα και νομικά ε, προβλήματα τι θα γίνει με τη νομική βάση, πώ θα προχωρήσουμε. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε και αυτά τα οποία είπαν αρκετέ συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και η κυρία Μπιλμπάο, είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ε, συμπεριληφθούν και άλλα πράγματα σε αυτό τον κατάλογο. Εάν το Συμβούλιο θέλει, ε, θα πρέπει να γίνει. Εγώ νομίζω ότι το Συμβούλιο, εάν του κάνουμε μια καλή πρόταση, δεν θα μπορέσει να την απορρίψει, διότι πώς θα εξηγήσει ε, την εχθρική του στάση το Συμβούλιο όταν μία γυναίκα στις τέσσερις στην Ευρώπη είναι θύμα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της ε, βίας, ε, κακομεταχείρισης. Ε, πώς μπορεί το Συμβούλιο να απορρίψει τα θέματα αυτά όταν υπάρχει ε, μια μακρά λωρίδα αίματος σε όλη την Ευρώπη που σημαίνει ότι κάθε μέρα σε όλη την Ευρώπη πεθαίνουν πάρα πολλές γυναίκες. Και γιατί, γιατί ίσως ο σύντροφός τους, ο σύζυγός τους, ο πρώην σύζυγός τους, ο ραβωνιαστικός τους, ο, ο άνθρωπος με τον οποίο συζούν λόγω ζήλιας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο τη σκοτώνουν. Νομίζω ότι το Συμβούλιο δεν θα μπορέσει να αποφύγει ε, το ενδεχόμενο να επιμηκυνθεί αυτός ο κατάλογος. Ε, θα πρέπει λοιπόν ενωμένε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση, διότι κατά την άποψή μου θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Θα φτάσουμε στις ευρωεκλογέ και θα μπορέσουμε να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες, κοιτάξτε, εμείς κάναμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, η κυρία Μαρζικέτη, θέλει το λόγο. Όχι. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σημειώνω την ενδιαφέρουσα νομική γνωμοδότηση. Προς το παρόν αυτό που μπορώ να κάνω είναι να αναφέρω αυτά που είπε και η Αντιπρόεδρος Τρέντινγκ στην προφορική ερώτηση που της έγινε το Φεβρουάριο. Πρόκειται για την ερώτηση 4 του 2013, όπου ανέφερε ότι όσο έχει σήμερα η νομοθεσία του άρθρου 83 παράγραφος 1 δεν επιτρέπει να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα ούτε για τον καθορισμό ούτε για τις κυρώσεις, ενδεχόμενες κυρώσεις για τη βία κατά των γυναικών. Προς το παρόν δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Αλλά βεβαίως ε, παρακαλουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τις εργασίες σας και θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε ε, σε αυτές. Και τώρα θα δώσω τη νομική υπηρεσία για να απαντήσετε και θα τελειώσουμε με την ησυχήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Συγήτρια, Ευχαριστούμε πολύ και όλα τα μέλη για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Πολύ σύντομα θα σας πω τι μας ζητήθηκε εμείς. Ποια είναι η αποστολή μας σαν νομική υπηρεσία. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας σαν αποτέλεσμα αυτής της νομικής γνωμοδότησης που υποβάλαμε βάσει της επιθυμίας της Επιτροπής σας βεβαίως. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε πολιτικό ρόλο. Εμείς είμαστε δεσμευμένοι, όπως λέει και το δικαστήριο, πρέπει να σας δώσουμε μια πραγματική κατάσταση και νομική γνωμοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν καλύπτει άλλα θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν. Εμείς ε, αυτή είναι η αποστολή μας, αυτό είναι το καθήκον μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε την πολιτική βούληση και επιθυμία αυτής της Επιτροπής. Πρόκειται απλώς για μια γνωμοδότηση και από πολιτικής απόψεως δεν δεσμεύει την Επιτροπή. Και καταλαβαίνετε, εγώ γνωρίζω την περιπλοκότητα και τη σοβαρότητα των υποθέσεων κακομεταχείρισης γυναικών. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να θεωρήσετε ότι προσπαθούμε να εμποδίσουμε την εργασία αυτής της Επιτροπής. Όπως πολύ σωστά είπαν τα μέλη της Επιτροπής, όντως προσπαθούμε να διερευνήσουμε ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει δράση νομική. Υπάρχει το θέμα της ομοφωνίας του Συμβουλίου, που βεβαίως θα διευρύνει το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, θα ήθελα να σας απαντήσω προσθέτοντας δύο ή τρία στοιχεία ακόμα, έτσι ώστε να μπορέσετε να προσανατολιστείτε. Η συνθήκη ορίζει ότι δεν πρόκειται για νομοθετική διαδικασία, πρόκειται για μια απόφαση του Συμβουλίου. Είναι ακριβώς όπως ε, όταν θέλουμε να υπάρξει μεταρρύθμιση της συνθήκης. Το Κοινοβούλιο βεβαίως μπορεί να κάνει μία πρόταση. Να υποβάλει πρόταση να γίνει κάτι τέτοιο. Και αν αυτή είναι η επιλογή σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας δύο σημαντικά στοιχεία που ορίζει η συνθήκη. Η διεύρυνση των, του καταλόγου των εγκλημάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σοβαρά εγκλήματα με διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να εξαρτάται είτε από τη φύση της αξιόπινης πράξης, είτε από την ανάγκη να υπάρξει μια διαφορετική νομική βάση. Αυτό ουσιαστικά μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς σαν επιχείρημα για να προσθεθεί η βία κατά των γυναικών στον κατάλογο των εγκλημάτων αυτών. Τώρα, μιλήσατε για την στατιστική πλευρά και τους άλλους τομείς. Όντως και αυτό μπορεί να ε, αποτελέσει ένα επιχείρημα υπέρ του να προσθέσουμε αυτά τα εγκλήματα στον κατάλογο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Οι άλλοι τομεί ε, σαφώς και μπορεί να αποτελέσουν ένα σοβαρό επιχείρημα. Η νομική μας νομοδότηση λαμβάνει υπόψη τους τους σημαντικούς αυτούς τομείς και την ε, ανάθεση εξουσιών. Μιλάμε για την αρμοδιότητα στο ποινικό δίκαιο, στις ποινικέ υποθέσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κοινοτικό δίκαιο ο νομοθέτης μπορεί να υιοθετήσει μέτρα για όλους τους τομείς του ποινικού δικαίου. Και αυτή είναι η κύρια, αν θέλετε, επιφύλαξή μας. Γι' αυτό και ο συνάδελφος, και εγώ βεβαίως, περιοριστήκαμε στη γνωμοδότηση αυτή τη δυνατότητα να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο όσον αφορά την διεύρυνση του καταλόγου. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει συμβεί πάντως στο παρελθόν. Αυτό είναι και η τελική μου παρατήρηση. Αν χρειάζεστε περαιτέρω γνωμοδότηση και ανάλυση, μπορείτε να μας το ζητήσετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, η κυρία Νικολά. Εγώ θέλω να κάνω δύο Η βία κατά, όπως ξέρετε, ενός ατόμου είναι genus proximus. Έτσι χαρακτηρίζεται. Και μπορεί λοιπόν κανείς να κατηγορηθεί με αυτόν τον τρόπο διαφορετικά από άλλες κατηγορίες εγκλημάτων και αξιόπνων πράξεων. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει λύση γιατί υπάρχουν και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στην συνθήκη. Ίσως θα μπορέσουμε λοιπόν να συνδέσουμε το κείμενο αυτό με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, εάν υπάρξει διάταξη για την βία κατά των γυναικών και το άρθρο 83 της συνθήκης. Είναι θέμα ερμηνείας. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται ή όχι. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων είναι ένα έγκλημα που υπόκειται στο 83 παράγραφος 1. Είναι τα λεγόμενα ευρωεγκλήματα. Και στην γνωμοδότησή μας αυτό μπορούμε να το συμπεριλάβουμε. Όμως για την, τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει νομική βάση. πρέπει να γίνεται σεβαστός ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί νομική βάση. Τέλος, θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Να έχω και άλλη μια ερώτηση διευκρινιστική προς την νομική υπηρεσία όσον αφορά τη διαδικασία για την πρωτοβουλία μας υποβολή αιτήματο στο Συμβούλιο για να υπάρξει προσθήκη στον κατάλογο αυτών των εγκλημάτων. Ποια είναι η διαδικασία σαν Επιτροπή και σαν Κοινοβούλιο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Επίσης, υπάρχουν ε, οκτώ κατηγορίες εγκλημάτων σε αυτόν τον κατάλογο. Εδώ πρόκειται για μια διαδικασία που χρειάζεται κύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια ή απλώς τροποποιείται ο κατάλογος κάτι που προϋποθέτει απλώς απόφαση του Συμβουλίου χωρίς κύρωση από τα, ευρωπαϊκά, από Εθνικά Κοινοβούλια. Η νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σαν να πρόκειται για τροποποίηση συνθήκης, αλλά η διαδικασία είναι απλούστερη. Δεν περνάμε δηλαδή από τα Εθνικά Κοινοβούλια, περνάμε από την λεγόμενη διαδικασία Παστρέλ, αλλά το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο δυσκολεύει τα πράγματα μόνο για τη Γερμανία. Αν θέλετε δεν υπάρχει διαδικασία κύρωσης όπως ε, για μια κανονική ε, τροποποίηση της συνθήκης. Όλα τα κράτη-μέλη, οι εκπρόσωποι αν θέλετε στο Συμβούλιο των Κατών Μελών πρέπει να εκφράσουν την ε, σύμφωνη γνώμη τους. Βεβαίως ο Γερμανός εκπρόσωπος θα ζητήσει την άδεια του Bundestag. Είναι εξαίρεση όμως η Γερμανία. Τώρα για τη διαδικασία. Ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου πρόταση. και η διαδικασία του άρθρου 225 δεν μπορεί να ισχύσει εδώ, γιατί ουσιαστικά η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να ζητήσει το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο. Μια έκθεση η οποία επισήμως δηλαδή στέλνεται στο Συμβούλιο. Ίσως όμως θα πρέπει να το επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο πριν σας δώσω μια τελική ε, απάντηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχουμε μόνο 18 λεπτά. Δύο εκθέσεις πριν την 12.30. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα επεξεργαστούμε εκ νέου το θέμα. Το σχέδιο έκθεσης και κατόπιν θα ακολουθήσει η υποβολή των τροπολογιών. Και τώρα περνάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση αξιολόγηση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Η συγκήτρια κυρία να αντικαθίσταται από την κυρία Γκαμπριέλα. Καταρχά, η κυρία Πιτικάινεν να ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να είναι εδώ για να παρουσιάσει την έκθεσή της σήμερα. Μου ανέθεσε μένα το καθήκον. Καταρχάς η συντάκτρια της γραμμοδότηση θα ήθελε να ε, τονίσει ότι η συμμεταχείριση είναι καθολική αξία και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρείται με κάθε τρόπο. Γι' αυτό ακριβώ και η συντάκτρια ε, θεωρεί ευπρόσδεκτη την αξιολόγηση του προγράμματος για την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων εγκλημάτων ε, και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα πιο ευάλωτα άτομα, δηλαδή τις γυναίκες και τα παιδιά. Πολλό δε μάλλον το γεγονό ότι οι γυναίκε πολλέ φορέ είναι θύματα πολλαπλών εγκλημάτων. Γι' αυτό ακριβώ μα υπενθυμίζει η συντάκτρια ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η συντάκτρια λυπάται διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει νομοθετικές πράξεις στον τομέα της βίας κατά των γυναικών, της ε, συμμετοχής ε, στην ε, πολιτική ζωή και την οδηγία για το θέμα του μισθολογικού χάσματος. Όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση θα πρέπει να κυρώσουν τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη για την προστασία και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και επαφείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ε, μέτρα για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωση το συντομότερο δυνατόν. Τέλος και κυρίως η εισηγήτρια θα ήθελε να υπενθυμίσει ε, το θέμα τη ε, ε, Ζητάτε να υπάρχει μία ευάλωτη προσέγγιση για τις γυναίκες, αυτό να αναφέρεται σε οποιαδήποτε επιμόρφωση και κατάρτιση του δικαστικού συστήματος και θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς ε, για τα θέματα αυτά ε, στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας να ε, επιληφθούν του ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε το λόγο, κύριε Μπιλμπάου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επειδή είμαι υπεύθυνη από πλευράς ε, της πολιτικής μου ομάδας, θα ήθελα απλώ να πω ότι έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ε, υπευλήθησαν αρκετές ε, τροπολογίες και θα αναλύσουμε την πρόταση που μας παρουσιάστηκε και θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε και την ανάγκη της περιφερειακής προοπτικής στην εξέλιξη του προγράμματος, διότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και κάποιους ε, άλλους τομείς πέραν των θεσμικών, να γνωρίζουμε και τι γίνεται ε, σε τοπικό επίπεδο για την ε, καταπολέμηση και της τρομοκρατίας και των οργανωμένων εγκλήματος. Ασχοληθήκαμε πολύ σήμερα με το θέμα της βίας κατά των γυναικών και τι γίνεται με την προστασία των θυμάτων τρομοκρατίας και θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε προτεραιότητα δεοντολογικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και να προσπαθήσουμε να υπάρχει πρόληψη αλλά και αποζημίωση στα θύματα. Ευπρόσδεκτα λοιπόν τα σημεία 4 και 5 της γνωμοδότησης και μία πτυχή που δεν έχει συμπεριληφθεί μεν αλλά ίσως θα έπρεπε είναι η δυνατότητα ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο καλύτερα και τις νέες τεχνολογίες στην εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης ε, για τις πτυχές τις οποίες προσπαθούμε να ενισχύσουμε. Πολύ ικανοποιητική λοιπόν η πρόταση και θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς με τη σειρά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μιλήσει. Ο εκπρόσωπος θέλει να κάνει κάποια προσθήκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά να πω ότι αυτή η γνωμοδότηση σχετίζεται με το σχέδιο έκθεση το οποίο παρουσιάστηκε από του επιτρεπέ ΑΦΚΟ και Γιούρι χθες. Υπάρχουν ορισμένα θέματα στην έκθεση αυτή τα οποία ε, αφορούν τις επιτροπές. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερο για αυτά, ε, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σχολιάσει ακόμα το σχέδιο έκθεση, ε, διότι το λάβαμε μόλι χθε και είναι προσωρινό προς το παρόν. Αυτό που θα θέλαμε από το Κοινοβούλιο είναι να έχει μία θετική αντιμετώπιση και να δει το τι μπορεί να γίνει μετά τη Στοκχόλμη, διότι λύγει το 2004, είναι ένα πρόγραμμα πενταετές, περιορισμένο λοιπόν όπως και τα προηγούμενα. Στο μεταξύ σε θεσμικό πλαίσιο τα προγράμματα αυτά <clears throat> έχουν αλλάξει, η πολιτική πλέον είναι ευρωπαϊκή και όχι εθνική το Κοινοβούλιο έχει ίσα δικαιώματα με το Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν αναμένεται το αντίκτυπο της γνώμης του Κοινοβουλίου να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα, προηγούμενα έτη. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει ανάγκη για τέτοια προγράμματα στο μέλλον, αν τα χρειαζόμαστε. Για το λόγο αυτό λοιπόν θα θέλαμε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δούνε αν είναι, αν έχει έρθει η ώρα να εξετάσουν καλύτερα τις ε, στρατηγικές τους για το μέλλον. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο που αναφέρθηκε εδώ, να σας πω ότι πληροφορίες από τους συναδέλφους μου που ασχολήθηκαν με αυτό είναι εξής. Δύο σημεία θα σας αναφέρω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει την πρωτοβουλία για δέσμευση, για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας από όλες τις μορφές βίας και βελτίωση των γνώσεων και της ε, συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων στα πλαίσια που μπορεί να δράσει. Μόλις μας είπε και η νομική υπηρεσία ότι δεν είναι εύκολο να βρεθεί η σωστή νομική βάση. Επίσης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ε, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση θα παραμείνουν προτεραιότητές μας Ήταν ε, αυτό μία από τις μεγάλες νομικές προτάσεις που έχουμε προτείνει το 2012 κάθετος 29 για την προστασία θυμάτων εγκλήματος. Αναφέρθηκε επίσης και η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας από τον Απρίλιο του 2011 η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση αυτή απαιτεί προηγουμένως λεπτομερή ανάλυση όλων των πολιτικών και των επιπτώσεών τους και ταυτόχρονα οποιαδήποτε πρόσθετη αξία που θα δώσει η προσχώρηση αυτή. Αυτό λοιπόν το έργο έχουμε αναλάβει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζουμε τα πάντα με λεπτομε... Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Συγητή, θα ήθελε να πει κάτι. Όχι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα σας πω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες 15 Ιουλίου. 12 το μεσημέρι, ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Κοινοβουλίου 18 Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών στις 3 Οκτωβρίου. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ελπίζω να προλάβουμε. Θα να ζητήσω την εισηγήτρια τώρα να προσπαθήσει στα 10 λεπτά που απομένουν, αλλά κυρία Γκαμπρέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι ήδη η έκθεση του κυρίου Τάνοκ ε, στην κατάσταση των, ε, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ είναι καλή έκθεση και εκεί λαμβάνονται υπόψη αρκετά σημεία που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών υπενθυμίζει την πρόκληση της ε, θνησιμότητας και των βρεφών ε, και των ε, γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης που είναι πολύ σημαντικές στην περιοχή και την πλήττουν την περιοχή, καλύτερη εκπαίδευση για τις γυναίκες και βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, επιμένει στην ανάγκη συμμετοχής των εκλογών και των γυναικών, κάνει έκκληση κατά του ακροτηριασμού γυναικών οργάνων, και ε, επισημαίνει ότι είναι κατεπίγουσα μεν η κατάσταση στο Μαλί, αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχουν και χρόνια ε, προβλήματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και ότι οι παραβιάσεις κατά των γυναικών ε, στην ε, περιοχή δεν αφορούν μόνο τις περιπτώσεις ενόπλης σύραξης. Επίσης, εμείς στη γνωμοδότησή μας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και για τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν προκειμένου στην περιοχή να ζήσουν κάποιες καλύτερες μέρες. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε στην πρόταση έκθεση να συμπεριληφθούν κάποια στοιχεία. Πρώτον, το γεγονό ότι οι γυναίκε μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο για την επίλυση των σειράξεων, θα πρέπει να βοηθήσουν για την ειρήνη στην περιοχή του Σαχέλ. Καμία χώρα δεν θα μπορέσει να προχωρήσει πολιτικά και οικονομικά εάν αφήσουμε στην άκρη και παραγωνίσουμε το 50% του πληθυσμού. Γι' αυτό ακριβώ και στη διάσκεψη που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση τον περασμένο Απρίλιο, με την κυρία Άστον και τον κύριο Ρωμάνο Πρόντι ε, τον οποίο υποστηρίζουμε για την πρωτοβουλία, ήρθαμε σε επαφή με χώρες ε, και οργανώσεις της περιοχής. Συνειδητοποιούμε ότι οι γυναίκες πρέπει να διαδραματίσουν πλήρη ρόλο στην προώθηση της δημοκρατίας και ακριβώς αυτό υπενθυμίζουμε και στη γνωμοδότηση. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και του Ευρωπαϊκού Οργάνου για την Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στον εξωτερικό τομέα τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικές Δράσεις θα πρέπει να ενθαρρύνει ώστε να λαμβάνονται νομοθετικά μέτρα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο συγκεκριμένα ε, τα οποία στόχο θα έχουν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών σε θέματα παιδείας, συμμετοχής ε, στον οικονομικό και πολιτικό βίο της χώρας. Τρίτον, η γνωμοδότηση επισημαίνει ότι πρέπει να μειωθεί η βία κατά των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών και είτε πρόκειται για άμεση βία είτε πρόκειται για αμέλεια σε περίπτωση νέων κοριτσιών. Και τέλος θα ήθελα να επανέλθω στην ε, περίπτωση του Μαλή και στη δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Διεθνούς Κοινότητας. Ε, καλωσορίζουμε την ε, διάσκεψη χορηγών για το Μαλή είχαμε συγκέντρωση άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν θα πρέπει αυτές οι υποσχέσεις να παραμείνουν κενό γράμμα και φυσικά τα κονδύλια δεν θα πρέπει να χρησιμεύσουν μόνο για στρατιωτικές ε, πτυχές. Θα πρέπει να χρησιμεύσουν και για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και για την προώθηση την πολιτική, της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής του συμμετοχής. Τέλος, η Επιτροπή Παρατήρηση των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της συμμετοχής των γυναικών στις εκλογές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω ότι η συνεισφορά μας στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα είναι πραγματικά σημαντική. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. ήθελα να αναφέρω και εγώ ορισμένα σημεία ακόμα, διότι η περιοχή αυτή μαστίζεται από ακραία φτώχεια και ένοπλε ε, συγκρούσεις, πολέμους και θα ήθελα λοιπόν να τονίσω την σημασία που έχει η συμμετοχή των ε, γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία, ιδιαίτερα σε διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με προηγούμενα ψηφίσματα που είχαμε. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω το ζήτημα της ατιμορρησίας, διότι δυστυχώς στην περιοχή αυτή διαπράττονται πολλά ποινικά αδικήματα, σεξουαλικά αδικήματα, εγκλήματα βίας και μαστίζεται το σύστημα από μεγάλη ατιμορρησία. Υπάρχουν ορισμένες ε, τροπολογίες αυτό, όμως σε γενικές γραμμές πιστεύω πως η έκθεση είναι εξισορροπημένη και θα συνεισφέρει θετικά στην έκθεση ΤΑΝΟΚ για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ, κύριο ε, Λαμπρίνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει το λόγο, δυστυχώς όχι για πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Γυναικών Πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό, η αναγνώριση του θετικού ρόλου στις ε, διαδικασίες διαβούλευσης στις τρίτες χώρες για την ε, δημοκρατία και τον δημοκρατικό και κοινοπολιτικό διάλογο. Και για το Μάλι αλλά και για την ε, όλη κρίση στο Σαχέλ έχουμε συγκεκριμένες δράσεις από μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Μαυριτανία αλλά και για το Μάλι. Πιο συγκεκριμένα 10 προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μάλι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ κυρίως για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή. Οι περισσότερες γυναίκες, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, της, τους τελευταίους μήνες συμμετείχαν και τα προγράμματα αυτά συνεχίστηκαν. Υπάρχει και το παρατηρητήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο στο Μάλι, αλλά και στο Τσάντ, στο, στην Πουρκίνα Φάσο και στην Βρυτανία. Μία παρατήρηση αντικειμενική, αμερόληπτη, συμπληρωματική με αυτή που γίνεται ε, μέσω της Αφρικανικής Ένωσης. Στη Μαυριτανία από το 2009 οι πρωτοβουλίες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ε, επικεντρωθεί σε τέσσερις άξονες. Υπάρχουν τέσσερα προγράμματα 500.000 ευρώ για την καταπολέμηση της δουλείας που πλήττει κυρίως τις γυναίκες, την πρόληψη ιδιαίτερα για γυναίκες και νέα κορίτσια που είναι θύματα βίας και θα ξεκινήσει και ένα νέο πρόγραμμα. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις για συμμετοχή στην Μαυριτανία. πολέμηση της δουλείας. Τώρα, για το 2011 και 2012 χρηματοδοτήσαμε με 4 εκατομμύρια ευρώ τέσσερα προγράμματα για τον ε, οικογενειακό προγραμμα... Ε, προγραμματισμό στην Ιγυρία το 2013 ξεκίνησε η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 200.000 ευρώ για την υποστήριξη πρωτοβουλειών στην κοινωνία των πολιτών και για τα σοφρονιστικά ιδρύματα, την εκπαίδευση, την ελευθερία έκφρασης και την ενημέρωση για τα ίσα δικαιώματα, πάντα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. Τέλος, Η Υπηρεσία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ξεκίνησε και μία πρωτοβουλία τέλος Ιουνίου θέτοντας προτεραιότητες όπως την καταπολέμηση των δολοφονιών παιδιών, κυρίως μικρά κορίτσια είναι θύματα αυτών των δολοφονικών πράξεων αλλά και ε, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα προγράμματα που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών. Η Να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες αυτές τις πολύ συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που στηρίζουν την ε, πρότασή μας και ελπίζω να φτάσουμε σε μια θετική πρόταση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες 15 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα είναι η προθεσμία. Θα ψηφίσουμε 2 Σεπτεμβρίου Νομίζω τελειώσαμε και με το σημείο 12. Και σας εύχομαι σε όλους καλή όρεξη.